Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Όλοι είναι εδώ, νομίζω, ε, που χρειάζεται για να ξεκινήσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 10 και 4 θα έχουμε την έκθεση του κυρίου Γκαρσία Ραμών, του κυρίου Γκαρσία Ραμών για τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική των καταναλωτών. Κάποιες μικρές ανακοινώσεις θα τις κάνω όταν έρθουν και άλλοι συνάδελφοι πριν τις ψηφοφορίες. Και μετά έχουμε κάποια τεχνικά θέματα για τα δασοκομικά μηχανήματα. So that's, that's the plan for this morning. Um, I'm very pleased um, uh, to welcome uh, Vivi Michou from από Justice. Uh, also we have... Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, τους Νίκ. Γενικά διάφορους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, προσπαθώ να πω τα ονόματα τώρα και δεν τα καταφέρνω. Έχουμε τον κύριο Νεοπτολέμου από, το, από την Προεδρία. ο οποίος προεδρεύει της ομάδας του Συμβουλίου για τα θέματα καταναλωτών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόταση. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία θέλουμε να προχωρήσει, γι' αυτό κάνουμε και έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και θα σχολιάσουμε αναλυτικότερα τις προτάσεις της Επιτροπής σε λίγο χρόνο. Θα ζητήσουμε από τον εισηγητή να μας πει προς ποιες κατευθύνσεις θέλει να προχωρήσει. Κύριε Γκαρσία Ραμόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάμε σήμερα με ναι, το έργο μας για αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από αυτό το σημαντικό θέμα αυτής της έκθεσης. Ε... Ξεκινώ λοιπόν λέγοντας αμέσως ότι πήρα την εντολή από αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή τον μήνα Ιούλιο για να ξεκινήσω με τη διατύπωση αυτής της έκθεσης σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ατζέντα θεματολόγια για τους Ευρωπαίους καταναλωτές για να προαθεί η εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη. Είναι αυτονόητο ότι κινούμε φυσικά από κάποια προηγούμενα αιτιολογικά ή ε, σκέψεις με προηγούμενα θέματα που έχουν συσσωρευτεί και συλλεχθεί στο μέτρο που αυτή η ατζέντα, το θεματολόγιο, στοχεύει να καθορίσει τα κυριότερα μέτρα τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την ικανότητα στους, ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση των καταναλωτών και να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη. Παράδειγμα. Για παράδειγμα έχουμε την έκθεση για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πράξη για την ενιαία εσωτερική αγορά, την ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο, την ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον οδικό χάρτη όσον αφορά την αποδοτικότητα, την πιο αποδοτική χρήση των πόρων μας. Όλα αυτά στοιχεία σε μια φαρέτρα, σε ένα σύνολο που αποτελούν μέρος και τμήμα των συζητήσεων και των θέσεων που υιοθετούμε και υιοθετήσαμε σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Στον χρονορίζοντα του προγράμματος τώρα για τον ορίζοντα 2020 στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την ε, θέση των καταναλωτών υπό μια άποψη λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα υγείας φυσικά, ασφάλειας και την αηφορία, τη βιωσιμότητα της μελλοντικής ανάπτυξης σε όλα αυτά στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε και να εξετάσουμε, να δούμε ότι αυτή η έκθεση που σήμερα θα συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή στα πρώτα της βήματα εντάσσεται, τοποθετείται σε ένα πολύ συγκεκριμένο εξειδικευμένο πλαίσιο συγκυριακά. Και αυτό είναι το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης σε αυτή τη συγκυρία και κοινωνικής κρίσης που περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα κάποιες από τις χώρες που την συναποτελούν. Θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος των καταναλωτών μέσα στο συνολικότερο οικονομικό και κοινωνικό ευρωπαϊκό σύστημα και να δούμε επίσης πώς αυτή η οικονομική συγκυρία έχει επιπτώσεις και επηρεάζει τους καταναλωτές. Ακριβώς σε σχέση με το κλίμα εμπιστοσύνης, την εμπιστοσύνη από πλευράς τους προς το οικονομικό σύστημα γενικότερα. Οι καταναλωτές μπορούμε να το δούμε ως εξή. Πρέπει, πιστεύω, να το προσεγγίσουμε όχι αυστηρά και αποκλειστικά ως ένα θέμα που αφορά την αγορά, αλλά το αντίθετο, ως ένα θέμα και αντικείμενο που αφορά το δίκαιο και τα δικαιώματα. δικαιώματα. Οι πολίτες πρέπει να είναι αντικείμενο δικαίου και να έχουν δικαιώματα, να έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας και με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους σε μια συγκεκριμένη στιγμή όπου η ανεργία, η μείωση θέσεων απασχόλησης, η αύξηση της ανεργίας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η συρρήκνωση, η μείωση της ιδιωτικής αποταμίευσης, η αύξηση των ανισοτήτων, όλα αυτά είναι πτυχές που συνδέονται και συγκλίνουν και συναρτώνται ώστε να αλλάζουν οι συνήθειες κατανάλωσης από πλευράς των καταναλωτών και το είδος και ο τρόπος κατανάλωσης σε αυτό το βαθμό μπορούμε να δούμε μια αλλαγή όλας των χαρακτηριστικών των καταναλωτών. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα την εντάξουμε και θα την ε, εμπλαισιώσουμε στην ε, έκθεση που θα συντάξουμε, που βρίσκεται υπό σύνταξη. Και ιδιαίτερα εδώ λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στις ανάγκες των πιο ευάλωτων καταναλωτών μέσα σε όλα αυτά. Και επίσης να δούμε την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι ενώσεις και σύλλογοι καταναλωτών που πολλές φορές ε, πλημμυρίζονται και τους ξεπερνούν τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε. Γενικότερα το σχήμα αυτό προσέγγισης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρότασή της μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αξιόλογο στοιχείο θα έλεγα για να μπορέσουμε να εντάξουμε τις εργασίες που πρέπει να, το έργο που πρέπει να καλύψουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ακόμα και αυτές, σε αυτόν τον προβληματισμό, αυτές τις σκέψεις που μόλις σας προανέφερα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα ιχνηλασιμότητας, ανείχνευσης, να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος σε συγκεκριμένες καταστάσεις όσον αφορά τις ετικέτες ε, στη συσκευασία προϊόντων και τους κοινωνικούς όρους υπό τους οποίους παράγονται αυτά τα προϊόντα περιβαλλοντική και κοινωνική αηφορία και βιωσιμότητα όσον αφορά την παραγωγή και τις υπηρεσίες ε, και όσον αφορά την εργασία γενικότερα. Και όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα συμπεριλάβουμε και να τα εξετάσουμε όπως πρέπει με τον σωστότερο τρόπο σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει επίσης να προβληματιστούμε και να αναφέρουμε, να πούμε κάτι για την κατάσταση των Ευρωπαίων καταναλωτών σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο που όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιείται και όπου οι εμπορικοί κανόνες και διατάξεις επηρεάζουν και τα αγαθά και τις υπηρεσίες πολυσχηδώς όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε και πολλές φορές και σε ευρύτερους τομείς όπως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ή σε άλλα πλαίσια. Πρέπει να δούμε πώς οι ρυθμίσεις των διεθνών αγορών για προϊόντα, για αγαθά και υπηρεσίες έχουν επιπτώσεις στους Ευρωπαίους καταναλωτές, πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη ζωή τους και κατά κάποιο τρόπο και η κρίση του χρηματοοικονομικού συστήματος σήμερα και οι αρνητικές επιπτώσεις που βιώνουν οι καταναλωτές σε κάποια οικονομικά προϊόντα, εξειδικευμένα οικονομικά προϊόντα που υφίστανται και για εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες δημιουργούνται πολύ ευάλωτες ε, καταστάσεις όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά θέματα. Για να αναφέρω την περίπτωση της Ισπανίας, όπου μυριάδες Ισπανοί αρνητικά επηρεάζονται όσον αφορά τα ποσοστά για την συμμετοχή και σε σχέση και με την ίδια την εργασία και που βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις από πλευρά των χρηματοοικονομικών θεμάτων στη ζωή τους. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εντάξουμε και να προσπαθήσουμε να τα εξετάσουμε στο σύνολο της έκθεσης, καθώς επίσης και τις πτυχές που αφορούν την υγεία και την εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση. Και για να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτή η έκθεση αυτό το θεματολόγιο, η ημερήσια διάταξη για τους καταναλωτές, πώς λέω, ποιες θα είναι οι οικονομικές διαστάσεις όλων αυτών, η οικονομική τους εμβέλεια, θα είναι, ποιο θα είναι το οικονομικό κόστος για να δρομολογηθούν και να ξεκινήσουν δράσεις. Πρέπει να κάνουμε κατά προσέγγιση μια εκτίμηση, να δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και οι πιθανότητες, οι εναλλακτικέ δυνατότητες για την υλοποίηση, την εφαρμογή όλων αυτών για να μην παραμείνουμε απλά στα λόγια, σε θεωρητικές δηλώσεις ρητορικές αλλά να είναι ένα πραγματικό μέσο, ένα πραγματικό εργαλείο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και οι καταναλωτές στο σύνολό τους να είναι ένα στοιχείο για να αναζωογονηθεί το οικονομικό σύστημα συνολικά υπό αυτές τις προοπτικές. Έτσι λοιπόν τούτων λεχθέντων θα ακούσω προσεκτικά, θα φουγκραστώ ποιες είναι οι απόψεις σας σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και είμαι φυσικά πρόθυμος και ανοιχτός όχι μόνο να ακούσω τις απόψεις και τα σχόλιά σας, αλλά να προσπαθήσω όλα αυτά να τα εντάξω και να τα συμπεριλάβω, ώστε στο τέλος να καταλήξουμε σε μια έκθεση που η δική μας κοινοβουλευτική θα πρέπει να συζητήσει και να εγκρίνει και που θα είναι η καλύτερη δυνατή. Σας ευχαριστώ. Uh, well, thank Σας ευχαριστούμε κύριε Γκαρσές Ραμόν. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αφετηρία για τη συζήτηση. Θα περάσουμε τώρα σε ένα γύρο ομιλιών των σκιωδών εισηγητών. Η κυρία Καλνιέτε απουσιάζει. Φαντάζομαι ο κύριος Βάπ θα αντικαταστήσει εκ μέρους του ΕΛΚ. Ο κύριος Σμιτ θα αντικαταστήσει τον κύριο Ροσφόρ. Η κυρία Ρούλε είναι παρούσα. Εγώ θα αναπληρώσω τον σκιώδη συγητή της δικής μου ομάδας. Ξέρω ότι θέλουν το λόγο η κυρία Σενάλοβα, η κυρία Χέντ. Θα δούμε. Ποιος θα ξεκινήσει, ο κύριος Φαπ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι η ευγένεια το απαιτεί και είναι θετικό γι' αυτό. Αν τώρα εγώ σε εκπρόσωπος της ομάδας του ΕΛΚ για την κυρία Κανιέτε η οποία δεν μπορεί να παραστεί. Δύο-τρία λόγια θα πω για λογαριασμό της. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για όσα είπε. Έχουμε εδώ μια πολύ φιλόδοξη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι γνωστό ότι κάποια κράτη-μέλη στο πλαίσιο και περιθώριο των δυνατοτήτων τους βρίσκονται που πολλές πάμπολες προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για την διάταξη των οικονομικών αγορών και την υλοποίησή τους, αλλά και πολλά άλλα τα δυσχεραίνουν. Γι' αυτό έχω κάποιες επιφυλάξεις, αν θα έπρεπε να ανοίξουμε έναν άλλο πίθο δαναείδων για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών με το φιλόδοξο, το, φιλόδοξο πνεύμα είναι αξιόλογο σε αυτή την έκθεση σίγουρα Συμφωνούμε και το τόνισε ο κύριος Προλαλή σας ότι η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική και τότε μόνο μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν έχει παιδεία, κατάρτιση, επιμόρφωση που θα κάνει τους εργαζόμενους να είναι οι καλύτεροι στο πεδίο τους. Και έτσι να προσπαθήσουμε λοιπόν από την Επιτροπή να ενισχύσουμε τις γνώσεις, να ενδυναμώσουμε τις γνώσεις των εργαζομένων με ένα μέσο, με ένα εργαλείο, θα το ε, κάνουμε αυτό θα πρέπει να το δούμε και να λαμβάνεται από η απόφαση από του ίδιου του καταναλωτέ. Ε, από πλευρά ουσία το υποστηρίζω αυτό σε εγχείρημα, αλλά στα κράτη-μέλη όλα αυτά πρέπει να δίνουν δυνατότητε ενό εφικτού πλαισίου, δυνατότητα πραγματικά να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να δράσουν και να μην τα ξεπερνούν τα κράτη-μέλη όλα αυτά και για τον ανταγωνισμό, για το καλύτερο προϊόν, στο τέλος τέλος πάλι θα πρέπει ο καταναλωτής να εγκρίνει ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα επιλέγει. Τούτων όλων λεχθέντων λοιπόν θα ήταν πολύ θετικό να αυτά τα λαμβάναμε έτσι υπόψη. Σε κάποια σημεία νομίζω θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω επ' αυτών. Θέλω μόνο να πω ότι αδειμονώ να δω Προσβλέπω να δω τι θα γίνει τώρα η Επιτροπή μάλλον, έχει κάποιες, ε, μάλλον κρατά κάποια χαρτιά στα χέρια που δεν έχει αποκαλύψει ακόμα σε σχέση με τις, ε, την διευθέτηση κάποιων ε, προβλημάτων όσον αφορά θέματα εργατικά ή απεργίας. Χαιρόμαστε και θέλουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η συζήτηση από πλευράς του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σμιτ, εκ μέρους του κυρίου Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φιλελεύθερη είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τον Ευρωπαίο Καταναλωτή, γιατί έτσι υπογραμμίζουμε ε, τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Για αυτήν την άποψη η ανακοίνωση κάνει μια καλή επισκόπηση των μέχρι τώρα επιτευγμάτων αλλά και της μελλοντική πορείας προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ε, εσωτερική αγορά να προστατευτούν και να βελτιωθούν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Είμαστε υπέρ του γενικού προσανατολισμού του κειμένου, τον θεωρούμε εξαιρετικό. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα μόνο σημεία. Πρώτον, συμφωνούμε με τι δράσει που, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2014 για να εξασφαλίσει ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων, ε, ιδιαίτερα με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για την ε, ασφάλεια των ε, προϊόντων. Επίσης έχουμε τον πράσινο χάρτη για την ασφάλεια πολλών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τους ευάλωτους καταναλωτές. Δεύτερον, θέλουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή της οδηγίας και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα των μέτρων αποζημίωσης. Τώρα εξετάσουμε και την οδηγία RDR για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών και το ODR ε, για την επιγραμμική επίλυση διαφορών. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικά νομοθετικά μέτρα για, την, ε, για τα ένδικα βοηθήματα των καταναλωτών. Εγώ είμαι υπέρ ε, συλλογικών προσφυγών, αλλά δεν είναι κρατούσα αυτή η γνώμη. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να αφυπνιστούν οι πολίτες ως προς τα δικαιώματα που έχουν ως καταναλωτές. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να βρούμε το σωστό τρόπο για να ενημερώσουμε σωστά και την κατάλληλη στιγμή τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα πρέπει οι καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους ε, σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον και για να μπορούν να τα ασκήσουν και αποτελεσματικά. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, ε, να χορηγήσουμε στους καταναλωτές ε, συγκρίσιμα, αξιόπιστα και προσπελάσιμα στοιχεία, ιδιαίτερα για τις διασυνοριακές περιπτώσεις. Θα πρέπει να τους βοηθούμε να συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές, αλλά και την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των αγαθών και των υπηρεσιών. Και ένας από τους τρόπους να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό είναι να αναπτύξουμε συγκρίσιμους ε, ιστοχώρους ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογραμμίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση, γιατί για τις καθημερινές αγορές προσφεύγουν στο διαδίκτυο οι καταναλωτές. Και έχουμε και το πρόγραμμα μέχρι το 2020 που εξετάζεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κοιτάσετε υπέρ της ανάπτυξης ε, τέτοιων ε, ιστοσελίδων, καθώς και τη θέσπιση δεοντολογικών κωδίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην είναι παραπλανητική ε, αυτή η στοχώρη για τους καταναλωτές. Ο κύριος Ροσφόρ προσβλέπει σε καρποφόρες συζητήσεις και σε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Η Χάιντι Ευχαριστώ. Και εμείς χαιρετίζουμε αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαιρόμαστε για τις ενδιαφέρουσες συζήτησεις, σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να επισημάνω και να πω ότι δεν πρέπει να υπάρξει επικάλυψη και διπλασιασμός έργου και εργασίας. Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν θα έπρεπε να αναμείνουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν στην έκθεση του κυρίου Ροσφόρ. Αν τα χρειαζόμαστε ή όχι πρέπει να προσέξουμε να μην διπλασιάζουμε πρωτοβουλίες και υπάρχει επικάλυψη. Είναι σημαντικό να δούμε προσεκτικά τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Γενική Οδηγία για την Παραγωγή Προϊόντων και για την εποπτεία και επόπτευση αγοράς. Δεν ωφελεί αν δεν λειτουργούν τα συστήματα εποπτείας αγοράς και δεν είναι αποτελεσματικά. Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή πάντα λέγαμε ότι δεν υπάρχουν τυποποιημένες διατάξεις ε, και προδιαγραφές όσον αφορά την εποπτεία, την επόπτευση αγορών. Θέλω να το τονίσω αυτό. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Εδώ και χρόνια έχει προαναγγείλει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέτος στο Single Act ε, για την κοινή αγορά, δηλαδή την νομική πράξη, την δεύτερη νομική πράξη για την ενιαία εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τις συλλογικές προσφυγές, collective redress, μάλιστα θα διεξαγάγουμε συζητήσεις γι' αυτό, αλλά πιο σημαντικό είναι να πω ότι έχω προσωπικά κάποιες επιφυλάξεις προσωπικά όσον αφορά το θέμα της πληροφόρησης και ενημέρωσης των καταναλωτών. Και όταν τώρα δούμε την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, καταδεικνύεται σαφώς ότι με μια πλημμυρίδα στοιχείων πληροφόρησης και πληροφοριακών στοιχείων δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ε, το καλό, το θετικό οι καταναλωτές. Έχουν προβλήματα, δεν είναι εξοικειωμένοι και καλά ε, εκπαιδευμένοι για να τα διηθήσουν όλα αυτά και να τα αντιληφθούν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσει αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί. Αλλά μόνο κάποιες, κάποια στρώματα, κάποιες κατηγορίες καταναλωτών βοηθά αυτό περισσότερο και όχι όλους τους καταναλωτές. Κρούω κόδωνα κινδύνου να μην ισοπεδώσουμε τα πράγματα σε σχέση με τους καταναλωτές. Εφόσον γίνεται αυτό εθελοντικά εντάξει, αλλά για την υποκατάσταση μιας καλής πολιτικής για τους καταναλωτές αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει να είναι στοχοθετημένο και δεν θα πρέπει να απαιτεί υπερβολικά πράγματα από τους καταναλωτές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ευχαριστώ. Σαν σκιώδης και εγώ να πάρω το λόγο για την πολιτική μου ομάδα. Θα ήθελα να μείνω σε αυτά που είπε η Χάιντι Ρούλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο κυκλοφόρησε κάποια ενδιαφέροντα κείμενα εργασίας για την βελτίωση της γνώσης και της ενημέρωσης του καταναλωτή. Ένας ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο στόχος και όπως ε, υπογράμμισε και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών, μερικές φορές ο καταναλωτής αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της πλημμυρίδας ενημέρωσης την οποία δέχεται. Θυμάμαι που είχαμε μια συνεδρίαση γύρω από αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Επιτροπής από την κυρία Μακάθιν. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των θεμάτων των καταναλωτών σε περιόδους δυσκολίας δημοσιονομικής πρέπει κυρίαρχα να είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρόσθεσης, αν θέλετε, αξίας στην προσπάθεια ενημέρωσης του καταναλωτή και σε σχέση με τις ροές της ενημέρωσης και σε σχέση με τις ροές της διασυνοριακής της ενημέρωσης Θέματα λοιπόν όπως η πληροφόρηση για θέματα ασφαλείας των προϊόντων, έλεγχη στις εισαγωγές, ψευδεπίγραφα προϊόντα, είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας. Θυμίζω ότι όπως είπε και ο εισηγητής ότι σε μία περίοδο όπου οι καταναλωτές έχουν περιορισμένους προϋπολογισμούς μπορεί να στραφούν σε ελκυστικά οικονομικά προϊόντα, τα οποία όμως να είναι χαμηλής ποιότητας ή και ψευδεπίγραφα. Πρέπει λοιπόν εμείς να φανούμε προσεκτικοί στα σχόλια που θα κάνουμε στην πρόταση, γιατί όσο περισσότερο μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε, θα δώσουμε και ουσία και βάρος στις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, τίθεται το θέμα της επιβολής των αποφάσεων. Έχουμε ε, μιλήσει και για την οδηγία για τις ε, μη νόμιμες εμπορικές πρακτικές ή στρεβλές εμπορικές πρακτικές. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Ξέρουμε ότι δεν εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο η οδηγία αυτή σε πολλές χώρες λόγω έλλειψης πόρων, λόγω ανυπαρξίας κατάλληλων μηχανισμών επιβολής και εφαρμογής των ρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να ενημερώσουμε τους καταναλωτές στον τομέα των δικαιωμάτων τους, να ξέρουν τι θα περιμένουν από τις ε, τοπικές καταναλωτικές οργανώσεις και από τις αρχές της χώρας τους. Δεν έχουμε χρήματα βέβαια για τεράστια πανευρωπαϊκά προγράμματα ή για νέους τρόπους πιστοποίησης λοιπά. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν πλέον. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν σωστές ας πούμε ιστοσελίδες για την ενημέρωση των καταναλωτών, να έχουν σημεία επαφής με τις καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες καλούνται εδώ να παίξουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο. Σχετικά με τα μελλοντικά προγράμματα. Το πακέτο, εν πάση περιπτώσει, για τις ταξιδιωτικές εμπορικές δραστηριότητες είναι κάτι ό,τι έχει σχέση με μετακινήσεις, ταξίδια κτλ. Είναι ένα πακέτο το οποίο προκαλεί κάποιες απορίες λόγω ε, της ε, σημαντικής ε, αλλαγής που υφίσταται η δραστηριότητα αυτή λόγω και της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτό άπτεται φυσικά και της οδηγίας για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπου και εκεί υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά τους καταναλωτές. Και στην ενέργεια επίσης πρέπει να κάνουμε πολλά για το κόστος της ενέργειας, την πρόσβαση και όλα αυτά είναι θέματα λοιπόν που άπτονται των καταναλωτών και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε στην πρότασή μας. Τελειώνοντας, να μιλήσω για, την, για τις δανειοδοτικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν κάποια, έχουμε ξεκαθαρίσει κάποιες απόψεις τις οποίες μπορούμε να προωθήσουμε. Να τελειώσω εδώ τώρα, σοβαρά θα τελειώσω. Έχουμε και άλλες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες γύρω από τα θέματα αυτά σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σε θέματα όπως σαν παράδειγμα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αν δείτε το scoreboard, τον πίνακα επιδόσεων, θα δείτε ότι είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ε, εμπορική δραστηριότητα, Υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα σε σχέση με ε, παράνομες εμπορικές, μη νόμιμες μάλλον εμπορικές πρακτικές, ε, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης κτλ. Εδώ τίθενται και κάποια δευτερεύοντα θέματα όπως το θέμα του τεχνικού ετήσιου ελέγχου, όπως το θέμα της εγγραφής εισαγωγικά των αυτοκινήτων από τη μία χώρα στην άλλη, όπως το θέμα της ε, αγοράς των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και πώς ελέγχεται. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες εδώ και να προσθέσουμε να, να, να εντάξουμε στο θέμα αυτό μία διάσταση προστασίας του καταναλωτή. Να βρούμε ένα σύστημα το οποίο σαν παράδειγμα να καταγράφει ε, ε, τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο και αυτό ε, λειτουργεί ε, στο Βέλγιο λέγεται Car και είναι κάτι το οποίο έχει μειώσει κατά πολύ τις απάτες ε, στον τομέα αυτό σχετικά με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει κάθε αυτοκίνητο. Μπορεί αυτό να είναι μια μορφή, μια υπηρεσία η οποία να μην είναι κερδοσκοπική και να μην επιβαρύνει πολύ την πρόταση. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω σήμερα. Ε, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι έχουν έλθει εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν θέλουν το λόγο. Η κυρία Σενάλοβα και μετά η κυρία Χέντα. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Η κυρία Σενάλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της και για την συζήτηση που έχουμε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα σχόλια της κυρίας Ρούλε και του Πρόεδρου. Σίγουρα θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας, αλλά και αφύπνιση του καταναλωτή. Και όταν μιλούμε για συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, ε, θα, δεν θα πρέπει μόνο να μιλούμε για σωστή ενημέρωση προκειμένου να κάνει περιστατωμένα την επιλογή του για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να εμπλέξουμε τους καταναλωτές στη χάραξη και διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών θα πρέπει να έχουμε πιο συχνές συζητήσει με εκπροσώπους των οργανώσεων καταναλωτών. Και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, και να καταστήσουμε πιο πρόσφορο το έδαφος για τις εργασίες τέτοιων οργανώσεων καταναλωτών. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωση σε πολύ περισσότερες γλώσσες για να μειωθεί κάπως το δημοκρατικό έλλειμμα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Συμφωνώ και με την κυρία Ρούλε ότι αυτή η ενημέρωση, η ενημερωτική εκστρατεία δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο για το Θεαθήνα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε ουσιαστικά τους καταναλωτές. Να τονίσουμε λοιπόν την ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τη σωστή εφαρμογή τους. Και ας μην ξεχνούμε και τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Εκεί αναφέρεται η ελπίδα για την υποβολή σύντομα πρότασης ό,τι αφορά τις συλλογικέ προσφυγές θα πρέπει και αυτό ο μηχανισμό να αποτελέσει ένα στο τμήμα τη πολιτική καταναλωτών. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό λοιπόν να θεσπιστούν σχετικά μέτρα. Ευχαριστούμε κυρία Σέναλοβα. Κυρία Χέτ. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εισαγωγή του. Και εγώ προσθέτω την φωνή μου απόλυτα και πλήρω στις σκέψεις που εξέφρασε ο ίδιος. Ακριβώς σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, χρηματοοικονομικής κρίσης, και όσον αφορά τους καταναλωτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εμείς στην Ευρώπη με τον καλύτερο τρόπο να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε οι καταναλωτές να τύχουν του υψηλότερου επίπεδου προστασίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό πάντα να καταβάλουμε αυτές τις προσπάθειες σε όλα τα θέματα καταναλωτών συνολικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε, να ελέγχουμε ότι οι κανόνες θα τηρούνται από όλους όσον αφορά το θέμα των συλλογικών προσφύγων. Συζητούμε αυτό το θέμα εδώ και τουλάχιστον 8 χρόνια. Όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκομαι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως επιτέλους. Ευάλωτοι η αδύναμοι οι καταναλωτές πρέπει περισσότερο να προστατεύονται και για νέους από διάφορες χώρες που συνάντησα σε μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε, μια μεγάλη σύναξη αντάμωση στις Βρυξέλλες. Οι νέοι αυτοί θεωρούσαν ότι ήταν επιζήμη αυτή η κατάσταση για αυτούς και συζητούσαν τις δυνατότητες να μπορέσουν να συμμετάσχουν για παράδειγμα οι βαρύκοοι σε αυτές τις ε, ε, δυνατότητες. Πρέπει να έχουν ειδικέ πληροφορίες οι βαρύκοοι και ε, να μπορούν να, όταν μετακινούνται για παράδειγμα με σιδηρόδρομο ή με άλλα μέσα να πληροφορούνται επαρκώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι αδύναμοι θα έλεγα μη προστατευόμενοι ευάλωτοι κανάλωτες και πρέπει να τους προστατέψουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο για το νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δύο Γενικών Διευθύνσεων. Και θα δώσω το λόγο και στον κύριο Νεπτολεμαίο από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Πρώτα κυρία Μισού, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ σήμερα εγώ είμαι στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, αλλά εκπροσωπώ και του συναδέλφους εδώ της ε, Γενικής Διεύθυνση ΣΑΜΚΟ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια μετά τη συζήτηση για τη νέα ατζέντα για τους καταναλωτές. Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε το Μάιο και σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Βέβαια σήμερα στις 10 θα αρχίσει η συζήτηση στο Λουξεμβούργο, στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού, για το θέμα αυτό του νέου θεματολογίου για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών. Φυσικά, όταν ε, οι δαπάνες για τους καταναλωτές είναι το 56% του ΑΕΠ, η ενεργό συμμετοχή ε, των καταναλωτών είναι θεμελιώδους σημασία για την ανάπτυξη και μάλιστα θα πρέπει συνειδητοποιημένοι, ε, συνειδητοποιημένοι καταναλωτές να συμμετέχουν σε αυτό και χαίρομαι για τη συμφωνία που εξέφρασαν ε, οι προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά αυτή την ε, αφύπνιση των καταναλωτών. Επίσης, θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει για μια περιεκτική, συνολική καταναλωτική πολιτική και εδώ και χρόνια εξετάζουμε τη μελλοντική μας πορεία. Εδώ προσπαθούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και διάλογο για να δούμε με τι νέα μέτρα μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την περσινή έκθεση Τριανταφυλλίδη, που ήταν πραγματικά πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Βέβαια, σήμερα που έχουμε μια σχετική πενία πόρων θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις μας με λιγότερα κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερο συντορισμό συνεργασία, ανταλλαγή εμπειριών και κοινέ δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμω, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα να εξασφαλίσουν ε, τους πόρους για τις εθνικές αρχές ε, εφαρμογής ε, ώστε να ανταπεξέλθουν και αυτές στην αποστολή τους. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσπαθούμε να ελέγξουμε όλο και καλύτερα την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και με το UCPD ε, προσπαθούμε με τους λίγους πόρους που έχουμε να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε και επίσης ε, συζητάμε με τα κράτη-μέλη την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών που ευελπιστούμε ότι θα ενσωματωθεί σε ένα μεστάξι προς τα τέλη του έτους. Το πρόγραμμά μα, η ατζέντα αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλιση πρόσβαση στου καταναλωτέ σε κατάλληλα 11 μέσα. Και οι προτάσει μα για το ADR και το ODR ε, έχουν θεμελιώδη σημασία για την υλοποίηση αυτού του δικαιώματο. Α μην ξεχνάμε κάτι που αναφέρατε και για τι οργανώσει των καταναλωτών. Μια ισχυρή φωνή των καταναλωτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική πολιτική για τους καταναλωτές. Η υποστήριξη λοιπόν από τις εθνικές κυβερνήσεις είναι απαραίτητη αν θέλουμε σωστή εφαρμογή αυτού, αυτού του προγράμματος. Και μάλιστα το νέο μας πρόγραμμα προτείνει ενισχυμένη ικανότητα αυτών των οργανώσεων καταναλωτών. Φυσικά χρειαζόμαστε μια υγιή, εύρωστη οικονομία και έντιμες επιχειρήσεις για να πατάξουμε τους αθέμητους εμπόρους, τους ε, εμπόρους που ασχολούνται με θέμητο ανταγωνισμό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ψηφιακή ατζέντα, τις μεταφορές, ε, την ασφάλεια των τροφίμων, που είναι κατά τη γνώμη των καταναλωτών οι σημαντικότερες πολιτικές ε, και οι πολιτικές με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον προπολογισμό των οικοκυριών. Και γι' αυτό θα στρέψουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στα θέματα αυτά. Α μην ξεχνούμε και τι δύο βασικέ προκλήσει που περιλαμβάνουμε στη νέα μα ατζέντα, προκειμένου να έχουμε πιο βιώσιμα σχήματα κατανάλωση και να προστατεύσουμε περισσότερο του ευάλωτε καταναλωτέ. Πολύ μεγάλη είναι η σημασία και των χρηματοπιστωτικών προγραμμάτων. Έχουμε βέβαια το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2014-2020, ένα τμήμα για τους καταναλωτές και ένα τμήμα για τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Θα συμβάλλουν και αυτά στην ε, υλοποίηση του θεματολογίου για τους καταναλωτές από το 2013 και μετά. Βέβαια αυτά τα δύο προγράμματα έχουν σχετικά μικρή ευέλεια, αλλά θα έχουν καταλητικό ρόλο για την ευρωπαϊκή πολιτική των καταναλωτών. Πιστεύουμε ότι αυτή, το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα των καταναλωτών δημιουργεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την κοινοτική πολιτική. Επίσης, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι το package travel, το πακέτο ε, για τα ταξίδια και τις υπηρεσίες αυτές θα ε, μπει στη διαδικασία αναθεώρησης για το 2013. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε τις προτεραιότητές σας. Ήταν σημαντικό για μας. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Τσίγκου. Ο κύριος Νεοπτολέμου από πλευρά Συμβουλίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω ακούσει με ιδιαίτερη ε, προσοχή τα όσα έχουν λεχθεί από τους προλαλήσαντες. Ε, να καλημερίσω όλους τους ε, παρεμπρεσκομένους από δικής μου πλευράς. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που λαμβάνω τον λόγο για να ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου για, τις, για το τι έχει πετύχει η Προεδρία στο θέμα του θεματολογίου των καταναλωτών, το οποίο βασικά θέτει εκείνες τις πολιτικές δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοθούν ε, από το κανονισμό, από το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει ενεξελίξη συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας στο Λουξεμβούργο αναφορικά με την υιοθέτηση συμπερασμάτων ε, στα οποία έχει ε, διαμορφώσει η Προεδρία και από αυτού θα ήθελα να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Μία μικρή παρέθεση να πω ότι η Προεδρία είναι αποφασισμένη και εκφράζει την πεποίθησή της ότι και το πρόγραμμα για τους καταναλωτές ο κανονισμός δηλαδή που θα χρηματοδοτήσει αυτές τις πολιτικές δράσεις που θέτονται στο θεματολόγιο των καταναλωτών βρίσκεται και αυτό ε, προς μια πολύ καλή πορεία και είμαστε πολύ ε, πεπισμένοι ότι θα, θα ολοκληρωθεί και αυτό πάρα πολύ σύντομα. Στο, ψήφισμα, το στο σχέδιο ψηφίσματος το οποίο έχουμε ετοιμάσει και όπως έχω πει συζητείται αυτή τη στιγμή στο Λουξεμβούργο εκφράζεται η ικανοποίηση για το θεματολόγιο των καταναλωτών και τους στόχους του οι οποίοι είναι η ενδυνάμωση της ασφάλειας των καταναλωτών όσον αφορά αγαθά υπηρεσίες και τρόφιμα μέσω της ενίσχυσης του κανονιστικού πλαισίου και της αποτελεσματικότερης υποπτίας της αγοράς. Η προαγωγή της γνώσης δεδομένης της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των αγορών, όπου οι καταναλωτές χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία και πληροφόρηση για να γνωρίζουν τα πάντα από το πραγματικό κόστος του καταναλωτικού δανείου έως την αρμόδια υπηρεσία παραπώνων τη βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας και την εξασφάλιση έννομης προστασίας, χωρίς τις οποίες δεν υπάρχουν δικαιώματα στην πράξη, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των σχετικών δικτύων επιβολής, την ευθυγράμμιση της πολιτικής προς τις κοινωνικές αλλαγές, προσαρμογή της πολιτικής στην καθημερινή ζωή με την προσαρμογή του δικαίου προστασίας των καταναλωτών στη ψηφιακή εποχή, αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές και μέρημνα για τις ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών όπως έχω ήδη ακούσει από τους προλαλήσαντες. Θέλω να δηλώσω κύριε Πρόεδρε ότι οι καταναλωτές είναι η κινητήρια δύναμη όπως έχει πει και η κυρία Μίχου προηγουμένως της οικονομίας και οι δαπάνες τους αντιπροσωπεύουν το 56% του αγαθάριστου χώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα του Συμβουλίου, επομένως, αναμένουμε να θεωρηθεί ως ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, πράγμα το οποίο θεωρούμε θεμελιώδες για την έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το σχέδιο το οποίο έχουμε ε, ετοιμάσει αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των αγορών και την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, ένας στους τέσσερις καταναλωτές δεν νιώθει αυτοπεποίθηση και ένας στους τρεις δεν ξέρει τα δικαιώματά του. Αναγνωρίζουμε ότι η αυτοπεποίθηση είναι βαρισίμαντη στο παρόν οικονομικό κλίμα. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η βελτίωση της νομοθεσίας που προστατεύει τους καταναλωτές είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αναγνωρίζουμε ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών θα πρέπει να ενδυναμωθεί όπως έχετε πει και εσείς προηγουμένως κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει η, σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις αυθύμητες εμπορικές πρακτικές. Πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των οργανώσεων, των καταναλωτών και να υποστηριχθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτέ και οι έμποροι περιορίζονται ακόμη στα εθνικά του σύνορα λόγω αδικαιολόγητων εμποδίων. Το θυματολόγιο για του καταναλωτέ απαιτεί συνεχή δέσμευση από την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην δύναμη των δικαιωμάτων τους. Στο σχέδιο ψηφίσματος το οποίο έχουμε ετοιμάσει κάνουμε αναφορά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Μαΐου του 2008 αναφορικά με την στρατηγική του καταναλωτή 2007-2013 κάνουμε αναφορά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Μαρτίου του 2010 για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Κάνουμε αναφορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου του 2010 αναφορικά με, την, ε, με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά. Κάνουμε αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου του 2011 όσον αφορά, θα το πω στα αγγλικά, relaunching of the single market. Και τέλος κάνουμε αναφορά στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου του 2012 αναφορικά με τη στρατηγική για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών. Οπομένω, η Προεδρία θεωρεί ότι μέσα από το επικείμενο ψήφισμα που πιστεύω ότι θα γίνει εντός των επόμενων λεπτών που μιλούμε. Δίδεται ένα σαφές και δυνατό πολιτικό μήνυμα ότι για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, για να προχωρήσουμε στην διέξοδο από την οικονομική κρίση, ο κεντρικός πυρήνας είναι ο καταναλωτής. Ελπίζω να ήμουν περιεκτικός, συγγνώμη που έχω ε, μακρογορήσει, αλλά χωρίς αδολεσχία κύριε Πρόεδρε, με ακρεφνή τρόπο, είναι αρίδηλο πλέον ότι ο καταναλωτής αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον μια τόσο επικαιροποιημένη έκθεση του Συμβουλίου για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ που προσήλθατε. Είσαστε ευπρόσδεκτοι και ασύνηθες στο τι προσήλθατε. Θα είναι πολύ χρήσιμο να διαβιβαστεί το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με το ψήφισμα, το σχέδιο ε, τώρα κατά πόσο θα γίνουν δεκτά από το Συμβούλιο, τουλάχιστον θα είναι χρήσιμο τα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εξοικειωθούν με αυτό. Σα ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά. Αυτό ολοκληρώνει αυτό το θέμα. Εκτό από το ότι θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκαρθία Ραμών να συνοψίσει αν θέλει και μετά το χρονοδιάγραμμα για το, το οποίο θα ακολουθήσουμε. Έχετε τον λόγο κύριε Γκαρθία Ραμών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις και σχόλιά τους σε αυτή την πρώτη συζήτηση. Επίσης ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο βέβαια για τα συμπληρωματικά στοιχεία πληροφορίας που, πληροφόρησης που μας έδωσαν και είμαι βέβαιος ότι θα ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Επίσης να πω ότι πρέπει να δούμε επαρκώς με τον σωστότερο τρόπο τις εκθέσεις ε, που ε, διατυπώνονται από το Συμβούλιο, από την Επιτροπή, την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και άλλα σώματα. Έχουμε ένα ολόκληρο σύνολο θεμάτων που μας δίνει την ευκαιρία για το θεματολόγιο για τους καταναλωτές να καταλήξουμε σε ένα σημαντικό μέσο, σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της στοχοθέτηση που αναφέραμε. Για το χρονοδιάγραμμα, σήμερα ξεκινήσαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με αυτή την εκκίνηση. Η πρόβλεψη Απρίλιο-Μάιο 2013 να είμαστε σε θέση αυτή η έκθεση να περάσει προς ψήφιση και έγκριση στην Ολομέλεια, στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειάς μας. Αλλά καθοδόν μέχρι τότε η ιδέα είναι στις 17 Δεκεμβρίου που θα έχουμε το πρώτο σχέδιο έκθεσης που θα κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, 17 Δεκεμβρίου λοιπόν, και με αυτή την ημερομηνία ως αφετηρία θα έχουμε ε, τη διαδικασία των τροπολογιών που θα ξεκινήσει με όλη τη γνωστή ε, διαδικασία και γνωρίζουν όλοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Θέλω να εκφράσω ρητά και κατηγορηματικά τη βούλησή μου ότι είμαι πρόθυμος και ανοιχτός σε όλα τα σχόλια ώστε να μπορέσουν και παρατηρήσεις ώστε να καταλήξουμε στο δυνατόν το πιο καρποφόρο εγχείρημα. Ευχαριστώ. Good. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε και λέμε ότι προσβλέπουμε να δούμε την έκθεσή σας. Έχετε μέχρι την 26η Νοεμβρίου να τα καταφέρετε να τα διατυπώσετε. 17 Δεκεμβρίου λοιπόν κατάθεση, 10 Ιανουαρίου κατάθεση τροπολογιών, εκπνέει προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών κατά τις ε, διακοπές των Χριστουγέννων θα προβληματιστούμε να δούμε τι θα γίνει. Θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Αυτό είναι το διευρυμένο χρονοδιάγραμμα. Θα μπορέσουμε έτσι να επικαιροποιήσουμε όλες τις πτυχές μέχρι τότε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ Συμβούλιο και Επιτροπή. Συνάδελφοι, κάπω καθυστερούμε χρονικά, αλλά νομίζω μπορούμε να καλύψουμε αυτή την ε, έλλειψη χρόνου, την διαφορά που έχουμε από το πρόγραμμά μας με τις εκλογές. Πρωτού περάσουμε στην ψήφιση, κάποιε ανακοινώσει από πλευράς μου. Λίγη ησυχία παρακαλώ, υπάρχει πολύ φασαρία στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω απλά κάτι στα μέλη, ότι νομίζω είχατε μια πρόσκληση από πλευρά του προγραμματός για την ε, εβδομάδα εκκίνησης ε, της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Στο 2Q2 στην αίθουσα αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε όλους όσους αναμενόντουσαν. Στις 10 θα ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση. Θα έχουμε μια εναρκτήρια συνεδρίαση όπου θα υποδεχθώ εξ ονόματος του Κοινοβουλίου τους προσκεκλημένους ε, κύριο Μπαρόζο. Ο κύριος Ντελόρ θα έρθει επίσης ως πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δώσει τις δικές του εκτιμήσεις Επίσης θα έχουμε και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τον κύριο Μάριο Μόντι. Με όλα αυτά θα ξεκινήσουμε. Μετά θα έχουμε μια συνεδρίαση για τα επιτεύγματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς όπου ο αντιπρόεδρος κύριος Λουί Γκρέκ και η Ρόζα θα συμμετάσχουν από κοινού με άλλους ε, εξέχοντες ομιλητές και τον Τζον Ντάλι. Μετά το γεύμα θα έχουμε τις προκλήσεις της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ε, ε, με τον κύριο Μπαρνιέ, τον Κύπριο ομόλογο και τον κύριο Σβάμπ. Μετά βραβεία για τους νέους γενεά ε, για τη νέα γενναία ο κύριος Μπαρνέο, συνάδελφος κύριος Πιτέλα στο τέλος θα κλείσει τη συνεδρία στις 5 η ώρα. Θα είναι λοιπόν μια εορταστική εκδήλωση με πάρα πολλές ε, ε, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τα μέλη και να παρίστανται. Και για το διαδίκτυο νομίζω ότι μια και έχουν όλες οι δυνατότητες εξαντληθεί θα μπορούσατε παρόλα αυτά αν θέλετε να παραστείτε να μπορέσετε να συμμετάσχετε βρίσκεται πίσω σας ο συνάδελφος δεν μπορώ να δω Ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι ευχαριστούμε Κάριν Γκέρμπο από πλευράς της ε, ε, δανέζικης κυβέρνησης θα επιστρέψει στην ε, Δανία. Είναι η τελευταία κοινοβουλευτική της ίσως συνεδρίαση. Θέλω να διαβιβαστούν οι καλύτερες ευχές μας σε εκείνη. Δύο τώρα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα, εκείνο που αφορά την τελική παρουσίαση Τη έκβασης του αποτελέσματος των τριμερών διαλόγων για δύο πολύ σημαντικά και τεχνικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκια επί των οποίων εργαζόμαστε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι και καλωσορίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν γνωρίζω ποιος θα παρέμβει εξ ονόματος της Επιτροπής. Η Μπάρμπαρα, εξ ονόματος της Επιτροπής. Πολύ καλά. Από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και καλωσορίζω την κυρία Μαρία Τσίγκου, ε, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου θα δώσω τον λόγο όταν θα έχουν παρουσιαστεί και τα δύο χαρτοφυλάκια, ώστε να μας δώσετε τις απόψεις σας συνοπτικά και για τα δύο αυτά θέματα. Θα ζητήσω λοιπόν από τους ε, εισηγητές να συνοψίσουν για σας την έκβαση αυτής της μακρόχρον, μακροχρόνιας και εργόδους, κοπιόδους ε, διαδικασίας σε διαδικασίες τριμερών διαλόγων. Θα θέλαμε επίσημα να έχουμε την έγκριση από πλευρά σας συνάδελφοι των δύο αυτών θέσεων στους τριμερείς διαλόγους που θα υποβληθούν στη συνέχεια στην Ολομέλεια, Ολομέλεια σε δύο εβδομάδες, στην Ολομέλεια περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου. Και για να το επιβεβαιώσουμε αυτό είχαμε και την επιστολή από το Συμβούλιο που επιβεβαίωνε ότι αν ενεκρίναμε εμείς θα ενέκριναν και εκείνοι από Ο κύριος Κοφεράτη από βράση του κύριου Παντσέρη για την πρώτη οδηγία. Ξεκινάμε λοιπόν. Με ποια σειρά θα τα πάρουμε λέει ο πρόεδρος. Ας ξεκινήσουμε με τους γεωργικούς ελκυστήρες, τα τρακτέρ πρώτα. Ο κύριος Κοφεράτη θα παρουσιάσει εξ ονόματος του εισηγητή κύριου Παντσέρη την θέση αυτή. Κύριε Κοφεράτη έχετε τον... Ευχαριστώ. Ζητά συγγνώμη ο συνάδελφος κ. Παντσέρη, αλλά δεν μπορεί να είναι παρόν. Είναι όμως πρόεδρος της αντιπροσωπείας της διακοινοβουλευτικής με τις χώρες Μαγκρέμπ και βρίσκεται σήμερα στην Τίνιδα. Μου ζήτησε λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους σκιώδης εισηγητές στην γραμματεία του Κοινοβουλίου και όλους όσους συνεισέφεραν στη συζήτηση και στην επίτευξη κάποιων στόχων οι οποίοι αρχικά φαίνονταν ιδιαίτερως μακρινοί αλλά νομίζω ότι εν πολλής έχουν επιτευχθεί. Να υπενθυμίσω ποια ήταν τα καταπροτεραιότητα θέματα της διαπραγμάτευσης. Περιλαμβάνονται στα άρθρα 7 και 8 σχετικά με την λειτουργική ασφάλεια Υπάρχει επίσης το 16 που αφορά την ε, πρόσβαση στην πληροφόρηση για την ε, επισκευή και συντήρηση και τέλος <clears throat> υπάρχουν οι εφαρμοστικές διατάξεις. Η συζήτηση για τα άρθρα 7 και 8 έκλεισε θετικά. Ήταν μια μακρόχρονη ευαίσθητη συζήτηση, ε, όχι όπως είναι συνήθως οι τεχνικές συζητήσεις. Παρόλα αυτά η τα συμπεράσματα νομίζω ότι ε, ήταν ικανοποιητικά γιατί καλύψαμε τις ανάγκες που υπήρχαν στον τομέα της λεγόμενης λειτουργικής ασφάλειας. Το ίδιο έγινε επίσης και σε σχέση με την λεγόμενη ε, εργασιακή, αν θέλετε, ασφάλεια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας δηλαδή των μηχανημάτων, έχει μεγάλη σημασία, διασφαλίσαμε την προστασία σαν παράδειγμα αντικειμένων ε, ή επίσης τις πτώσεις ε, των οδηγών ή χειριστών μάλλον, μια ολόκληρη τεχνική προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Αυτά που είπα για το 7 και 8 ισχύουν και για το 16. Η συμβιβαστική λύση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα αυτού, δίδοντας σχετικές εγγυήσεις για την πρόσβαση σε διαδικασίες κατάρτισης και για τους εισαγωγικά εγκεκριμένους πιστοποιημένους επισκευαστές τεχνικούς αλλά και για τους ανεξάρτητους τεχνικούς και επίσης λαμβάνουμε υπόψη και τα ειδικά χαρακτηριστικά των λεγόμενων μικρών σειρών παραγωγής, κάτι το οποίο τεχνικά παρουσιάζει δυσκολίες. Τώρα, σχετικά με το πότε θα τεθεί σε λειτουργία, σε ισχύ, λάβαμε υπόψη τις επιθυμίες των συναδέλφων, την προσπάθεια να δημιουργηθεί δηλαδή μία θέση σε ισχύ σταδιακή, με διαφοροποιημένο χρόνο για τα νέα προϊόντα και τα πρωτότυπα έτσι ώστε από τη μία να επιβεβαιωθεί η αρχική ημερομηνία θέση σε ισχύ του κανονισμού και από την άλλη να υπάρξουν κάποια επιμέρους στοιχεία ευελιξίας τα οποία ζητήθηκαν. Γι' αυτό ακριβώς και λόγω του προβλήματος χρόνου που έχουμε <clears throat> Ο κύριος Παντσέρη θεωρεί ότι η πρόταση είναι καλή και θεωρεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να, από την Επιτροπή μας να υποστηρίξει την πρότασή του στα πλαίσια της ψηφοφορίας που θα γίνει σε λίγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ ε, ενημερωτική αυτή η σύνοψη για τα επιτεύγματα της διαπραγματευτικής ομάδας. Σκιώδη ήταν Σβάμπα, Ρούλε, μάντερ, υποφαινόμενο ε, Σαντίνη. Θέλει κανεί ε, από του Σκιώδη το λόγο? Όχι. Θα ψηφίσουμε αργότερα, αφού ακούσουμε όμω του εκπροσώπου του Συμβουλίου και τη Επιτροπή Τώρα θα μα παρουσιάσει ο κ. Βαντενκάπ τη δική του πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω και εγώ τα αποτελέσματα μετά τον Ιταλό συνάδελφο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους από τα τρία θεσμικά όργανα με βοήθησαν τα τελευταία δυόμιση χρόνια γιατί ανέλαβα το Νοέμβριο τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας στο έργο μου. Στη συνέχεια συνεργαστήκα με, με τις διαδοχικές προεδρίες, ε, Ουγγρική, Πολωνική, Κυπριακή. Ήταν πολύ ευρωπαϊκή αυτή η εμπειρία. Οι σκιώδεις ηγητές, ε, οι μάλλον σκιώδεις ηγήτριες, ε, οι κυρίες Βέστφαλ και Ρούλε, με βοήθησαν να εξοικειωθώ ε, και με την γερμανική μεθοδικότητα και να καταλήξουμε σε πολύ πιο ασφαλή μέτρα στον κανονισμό αυτό και ένα κλάδο ε, δικύκλων πολύ πιο βιώσιμο, πολύ πιο φιλοπεριβαλλοντικό στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε μόνο για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά κάποια πλονεκτήματα. Θέλουμε η κατάσταση να βελτιωθεί στην παγκόσμια αγορά και οι συνάδελφοι από τη Κίνα και την Κορέα θα πρέπει να τηρήσουν και αυτοί τις διατάξεις του κανονισμού, ώστε η δική μας βιομηχανία δικύκλων να έχει αρκετό χρόνο ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες διατάξεις. Ένα ε, θέμα επίμαχο ήταν τα συστήματα πέδησης για τις μοτοσικλέτες και βέβαια ως και όδηση, γιατί ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενεργό συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιμο για μας ε, αυτή η πολύ δραστήρια συμμετοχή του Προέδρου. Τώρα θα γίνει και μία μελέτη κόστους ωφέλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ε, εφαρμοστούν τα συστήματα αντιεπλοκής των τροχών για κάτω 125 κυβικών. Επίσης είπαμε ότι οι μοτοσυκλέτες ε, και ε, οι δίκυκλες και τρίκλες μοτοσυκλέτες ε, δεν μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διατάξεις, γιατί στα άρθρα 18 έχουμε πιο συγκεκριμένες διατάξεις για τη δυνατότητα αυτή. Επίσης έχουμε και τους ελέγχους βιωσιμότητας και αντοχής η Κομισιόν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 θα πρέπει να προβεί σε μια πιο διεξοδική ανάλυση για, για το Euro 5 και τα διάφορα είδη εκπομπών καυσαερίων. Σίγουρα οι κινητήρες αυτών των οχημάτων θα γίνουν πιο φιλοπεριβαλλοντικοί και έχουμε και τους κανόνες 4 και 5 για τους ισχυρότερους κινητήρες, ενώ για τα σκούτερ που ρηπαίνουν ιδιαίτερα, ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Euro 3. Σε συνεννόηση με τον κύριο Παντσέρη καταλήξαμε σε πολύ καλές συμφωνίες για τα οχήματα αυτά Βέβαια μπορεί να, να έχουν μείνει κάποιες αδυναμίες, αλλά πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε στη συνεργασία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε ένα αίσιο αποτέλεσμα και ο κλάδος έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες διατάξεις γιατί η θέση ισχύει ε, γίνει από την 1η Πρώτου του 2016 και όχι από το 2014. Και εγώ που είμαι μηχανόβιος ξέρω ότι η περίοδος αυτή είναι αρκετά μακροχρόνια, αλλά για τη βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρκετά μεγάλη μεταβατική περίοδος. Και με τον τριμερή διάλογο καταφέραμε να διεκπεράσουμε το θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε κύριε Βαντερκάμπ και για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίσατε στην υπόθεση αυτή. Το γεγονό ότι συνέπεσε η ιδιότητα του Προέδρου με του και όδους γιατί δεν νομίζω ότι ε, περιόρισε καθόλου κύριε Βαντερκάμπ. Δεν ξέρω, κυρία Ρούλε, κανένα άλλο από του σκιώδους ηγητέ. Όχι. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Μπάρμπαρα Μπομβισούτο που παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή όλους του τριμερείς διαλόγους και μετά στους εκπροσώπους του Συμβουλίου, της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου ε, και κυρίως στην κυρία Τσίγκου για να μας κάνει ένα σχολιασμό και κατόπιν θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Κυρία Μποβισούτο, καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο εισηγητές, τον κύριο Παντσέρη, τον κύριο Βανταρκάμπ, τον πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, του και ηγητές, τη γραμματεία της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και φυσικά και την Προεδρία για την πολύ καλή προσπάθεια και την άοκνη προσπάθεια που κατέβαλε για το πολύ τεχνικό και περίπλοκο αυτό θέμα που θα αποφέρει όμως τεράστιους καρπούς και πλονεκτήματα για το περιβάλλον, την ασφάλεια και για τους πολίτες γενικά. Πιστεύω ότι πραγματικά καταλήξαμε σε πολύ θετική και ισορροπημένη συμβαστική πρόταση. Τα πιο επίμαχα σημεία που μας επισήμαναν οι κύριοι Κοφεράτη και Βαντερκάμ καταφέραμε να διαθετηθούν και πιστεύω ότι το τελικό κείμενο και για τις δύο προτάσεις είναι πολύ θετικό και πολύ φιλόδοξο και από περιβαλλοντική άποψη και από άποψη ε, προστασίας και ασφάλειας ενώ ταυτόχρονα προβλέπουμε αρκετά μεγάλες μεταβατικές περιόδους για τους κατασκευαστές. Υπάρχει μια προσπάθεια και απλούστευση των διατάξεων προς όφελος ε, και των ε, επιχειρηματιών και των αρχών, των αρμόδιων αρχών αλλά έχουμε προβλέψει και κάποιες διαδικασίες ε, συντήρησης προς όφελος των πολιτών, αλλά και διαδικασίες ε, επίβλεψης της αγοράς. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα και ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του. Σας ευχαριστώ. Ο Φιλίπ Ζω, που ήταν επικεφαλής της ομάδας, θα ήθελα ε, να τον ευχαριστήσουμε θερμά επίσης. Και τελικός λόγος στην κυρία Τσίγκου εκ μέρους του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συγητές, μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής, ε, δύο μακρά δυόμιση χρόνια εξαντλητικών συζητήσεων απαιτήθηκαν στο Συμβουλίο αλλά τελικά τα καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μαζί σας. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η μεγάλη χρονική διάρκεια σε μεγάλο βαθμό φιλόταν στο Συμβούλιο, το οποίο ήθελε να προσαρμόσει και σε αυτές τις δύο προτάσεις και να μπορέσει να το κάνει αυτό με το βέλτιστο τρόπο όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες. Οι εισηγητές σας και οι σκιώδεις εισηγητές ευθύς εξ αρχής κατέδειξαν την προθυμία τους να προχωρήσουν στις επαφές με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντωμεταξύ δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή τοποθετήθηκε με ένα πολύ θετικό επικοδομητικό πνεύμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλίζονται αμφωτέρωθεν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών και των βιομηχανιών, όπως ε, ήδη θα γνωρίζετε, ο κανονισμός για τους γεωργικούς ε, ελκυστήρες ομόφωνα εγκρίθηκε στην Κορεπέρ καθώς επίσης σε σχέση με τον κανονισμό για τις μοτοσυκλέτες μόνο ένα κράτος μέλος ε, επισήμανε ότι θα πήχε και αυτό οφείλεται μάλλον σε μια γενικότερη επιφύλαξη και μάλιστα είπαν ότι θα καλωσόριζαν για τα δίτροχα και τρίτροχα και τετράτροχα τον κανονισμό. Αυτό τι αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι επιτύχαμε αναβαθμισμένη υψηλού επίπεδου ποιότητα σε αυτές τις συμφωνίες και ε, με, την υψηλή ποιότητα των τροπολογιών που καταθέσατε και έτυχαν διαπραγμάτευσης ε, πετύχαμε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο. Θέλω να τονίσω ότι το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα επετέφθη σε δύο πολύ περίπλοκα τεχνικού χαρακτήρα κείμενα και είναι πραγματικά στεναρή η πεποίθησή μου ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε δύο πολύ χρήσιμους κανονισμούς για το πλαίσιο το οποίο θα ισχύει κατά το επόμενο διάστημα για την προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, την ε, βιομηχανική καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Εξ όνομα του Συμβουλίου λοιπόν, όχι μόνο εξ ονόματος της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά όπως και αναφέρθηκε επίσης ε, εξ ονόματος όλων των προεδριών που συνεργάστηκαν για αυτό το χαρτοφυλάκιο θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, τον κύριο Παντσέρη και τον κύριο Φαντεκάμπ για τις εκθέσεις τους και την θετική συνεργασία που είχαν μαζί μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τον πρόεδρο της δικής σας κοινοβουλευτικής επιτροπής, τον κύριο Χάμπορ, για την διοργάνωση ενός πολύ γόνιμου, ε, πολύ γόνιμων τριμερών διαλόγων, αλλά επίσης και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διευκρινήσεις σε τεχνικού χαρακτήρα θέματα που έδωσε και επίσης ε, συνεχίζει να παρέχει κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών και επίσης την γραμματεία της ΣΥΜΚΟ για το έργο που επετεύθη καθώς επίσης ε, και για τους ε, τετράστιλους πίνακες σύγκρισης. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία του Συμβουλίου που μας υποστήριξε σε αυτό το εγχείρημα και προσβλέπω σε θετική υπερψήφιση αποδοχή από πλευρά σας και για τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και πάλι. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας παρουσιάσατε αυτές τις απόψεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το τεράστιο έργο που γίνεται ε, πέραν το φως, πέραν, μακριά από το φως της δημοσιότητας, γιατί πραγματικά αυτά τα δυόμιση χρόνια είχαμε πολύ εντατικές και άκρες προσπάθειες και σας ευχαριστώ που ε, αναφερθήκατε και στη γραμματεία μας. Θα ήθελα να επενέσω και το έργο των ε, επιτελείων των διαφόρων πολιτικών ομάδων και φυσικά τους εισηγητές μας πρώτα απ' όλα. Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτα για το κείμενο την έκθεση Παντσέρη. Θα ήθελα να κάνουμε πρώτα ε, έναν έλεγχο, αν έχετε όλοι τις κάρτες σας, ε, για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα έγκριση του κανονισμού για τους ελκυστήρες, έγκριση τύπου για τα οχήματα γεωργίας και δασοκομείας. Δασικά και γεωργικά οχήματα. Έχετε όλοι οι χριστιανοδημοκράτες τις κάρτες σας. Mr. is Mrs. Rura. Okay. We still have we still have uh, five people who've Πέντε, ακόμα έχουν κάρτες αλλά δεν ψήφισαν. Μήπως δεν δουλεύει το σύστημα, αναρωτιέται ο πρόεδρος. 31 υπέρ, κανείς κατά, μία αποχή. Λοιπόν, έγιναν δεκτές αυτές οι προτάσεις. Περνάμε στον κανονισμό για τις ε, μοτοσυκλέτες. Τύπους έγκρισης, έλεγχος αγοράς. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 33 υπέρ. Γιατί έχουμε δύο χωρίς κάρτες. Κανείς κατά μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Χειροκροτούμε και τους δύο εισηγητές λοιπόν. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία μας για τις υπόλοιπες εκθέσεις, δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας. Η πρώτη αφορά την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενίας αγοράς. Ο κύριος Αρίας Ετσεβερία είναι ο εισηγητής μας. Θέλετε να πείτε κάτι. Θα ξεκινήσω με την 22. Guard. Ποιο είναι υπεύθυνο για την ψηφοφορία σοσιαλδημοκράτε σήμερα, κυρία Σέλντερ Μόζε. Απλά να ξέρω σε ποιον θα αναφερθώ ε, για τις ηλεκτρονικέ ψηφοφορίες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ησυχία παρακαλώ. 26 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Προφορική 2. Αρία σε τσεβερία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συνεχίζουμε με την 31. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πολιτισμού 13. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Βιομηχανία 20 υπέρ κατά δεκτή. Πολιτισμός 14. Ηλεκτρονική ψήφος. 17 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. 33. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 34. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 35. Μακλάρκιν υπέρ. Κατά. Δεκτή. 37. Γκούσταυσον υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Προσθήκη στην 6 υπέρ κατά, δεκτή. Πολιτισμός 1 υπέρ, κατά, δεκτή. 38 υπέρ, κατά, δεκτή. Βιομηχανία 8 υπέρ, κατά, δεκτή. Βιομηχανία 10 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, δεκτή. 41 υπέρ κατά δεκτή. 43 υπέρ κατά απορρίπτεται. 42 κάμπο υπέρ κατά δεκτή. Βιομηχανία 33 υπέρ κατά δεκτή. 44 Γκάρντ υπέρ κατά Απορρίπτεται. Πολιτισμός 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Βιομηχανία 34 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Βιομηχανία 35 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 49. Κορέα Ντεκάμπος υπέρ. Κατά. Δεκτή. 50 build υπέρ κατά, δεκτή. 51 Μακλάρκινγκ. υπέρ, κατά, δεκτή. 52 Λόκεγκαντ υπέρ, κατά, δεκτή. 53 Μακλάρκινγκ. υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 64. Γκαλό υπέρ κατά δεκτή. Νομική 5 υπέρ κατά δεκτή. Νομική 6 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική για την νομική 6. Η κυρία Ρούλα είναι κατά. Τέλος της ψηφοφορίας δεν γίνεται δεκτή. 21 κατά 14 υπέρ. Πολιτισμός 18 υπέρ κατά Τοπολογία 65 υπέρ κατά δεκτή. 66 υπέρ κατά δεκτή. 67 υπέρ κατά δεκτή. 68 Άρχεται η ψηφοφορία για την 68. Πέρα της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 21 κατά απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν τώρα στην 69. Προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 18 κατά. Δεν γίνεται δεκτή. 70 υπέρ, κατά. Δεκτή. Η βιομηχανία 36 υπέρ κατά δεκτή. 71 υπέρ κατά δεκτή. 72 υπέρ κατά δεκτή. 73 υπέρ κατά δεκτή. 75 προσθήκη υπέρ κατά δεκτή. 74 γκρεκ υπέρ κατά δεκτή. Νομική 7 υπέρ κατά δεκτή, νομική 8 υπέρ κατά δεκτή, βιομηχανία 12 υπέρ κατά δεκτή, 76 υπέρ κατά δεκτή, νομική 9 υπέρ κατά δεκτή, νομική 10 προσθήκη υπέρ κατά δεκτή, συμβιβαστική 7 υπέρ κατά δεκτή. Βιομηχανία 18 προσθήκη υπέρ κατά δεκτή. Βιομηχανία 24 υπέρ κατά δεκτή. 83 λογρίπ υπέρ κατά δεκτή. Πολιτισμός 7 υπέρ κατά δεκτή. Πολιτισμός 3 υπέρ κατά δεκτή. Μπορούμε να δεχθούμε τις ε, τροπολογίες αυτές ομαδικά. Είμαστε στον πολιτισμό 4, 8, 12 νομική και πολιτισμός 11 μαζί παρακαλώ. Όχι, όχι. Ξεχωριστά λοιπόν. Πολιτισμός 4 υπέρ κατά δεκτή. Πολιτισμός 8 υπέρ κατά δεκτή. Νομική 12 υπέρ κατά δεκτή. Πολιτισμός 11 υπέρ κατά δεκτή. 84 Σβάμπ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Κυρία Ρούλε κατά 18 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία Μακλάρκιν προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 85 ψηφίζεται. η κυρία Ρόλα είναι υπέρ 18 ή υπέρ 15 κατά. Νομική 4. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. 19 υπέρ 15 κατά δεκτή. Πολιτισμός 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 86 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 86 παρακαλώ. Η κυρία Ρούλα είναι υπέρ. 24 υπέρ 11 κατά. 87 υπέρ κατά δεκτή. 88 υπέρ κατά δεκτή. 90 υπέρ κατά δεκτή. 89 έχει, είναι ταυτόσημη. 91 υπέρ κατά δεκτή. 93 υπέρ κατά δεκτή. 92 προσθήκη υπέρ, κατά, δεκτή. Βιομηχανία 19 υπέρ, κατά, δεκτή. Πολιτισμός 5 και 6 υπέρ, κατά, δεκτές. Νομική 1 υπέρ, κατά, δεκτή. 96 υπέρ, κατά, δεκτή. 94 προσθήκη υπέρ, κατά, δεκτή. 95 υπέρ, κατά, δεκτή. 97 προσθήκη υπέρ, κατά, δεκτή. Βιομηχανία 11 υπέρ, κατά, δεκτή. Νομική 13 υπέρ, κατά, δεκτή. 98 έξτρον Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 98. Πέρας ψηφοφορία. 13 υπέρ 21 εναντίον απορρίφθηκε. Πολιτισμού 16 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 17 πολιτισμός προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην ε, βιομηχανία 37 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίθηκε. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πολιτισμού 10 και πολιτισμού 12. Από κοινού 10 και 12. 10 και 12 υπέρ κατά εγκρίθηκαν, εγκρίθηκαν οι 102 του κυρίου Τρασκόφσκι υπέρ της 100. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 102. Είναι υπέρ η κυρία Ρούλε. Πέρας ψηφοφορίες Δύο δεν ψήφισαν ακόμα. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ, 15 εναντίον. Τροπολογία 103 του κυρίου Έγκστρομ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Βιομηχανίες 5 και 6. Από κοινού, εντάξει, ωραία, από κοινού υπέρ, παρακαλώ, 5 και 6 κατά εγκρίθηκαν και οι δύο. Τροπολογία 104 της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Νομικής, νομικής Επιτροπής 14 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 105 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 106 υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Η 107 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Να πάρουμε από κοινού τη ΣΥΤΡΕ 1 και 2 γίνεται εντάξει. Βιομηχανίας λοιπόν 1 και 2 από κοινού υπέρ κατά εγκρίθηκαν. Η επόμενη ομάδα στην παράγραφο 27 από κοινού της Πολιτιστικής Επιτροπής 2, Βιομηχανίας 7, 9 και 21 από κοινού υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν όλες αυτές. Παράγραφο 31 ε, και 32 υπέρ κατά εγκρίθηκαν. 27, 28, 29, 30 της βιομηχανίας υπέρ κατά εγκρίθηκαν. 27, 28, 29, 30. Παράγραφος 29. Τροπολογία 108 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 109 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίθηκε. Της νομικής επιτροπής 11 καλύπτεται ήδη. Νομίζω την επόμενη κατηγορία της Επιτροπής Βιομηχανίας να την πάρουμε από κοινού 17, 22, 23, 25 και 26. Όλες υπέρ, παρακαλώ, κατά εγκρίθηκαν όλες. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, απορρίφθηκε, είναι σαφές. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τώρα τις βιομηχανίες 3 και 4 από κοινού υπέρ, κατά, εγκρίθηκαν. Βιομηχανίες 16 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 της βιομηχανίας υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογίες 10, 11 και 12 από κοινού γίνεται εντάξει όλες στην ίδια αιτιολογική σκέψη. 10, 11, 12 υπέρ, κατά εγκρίθηκαν όλες αυτές. Τοπολογία 13 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τοπολογία 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τοπολογία 15 και 16 από κοινού γίνεται. Εντάξει, υπέρ 15 και 16 κατά εγκρίθηκαν. Αιτιολογική σκέψη σίγμα τάφα, τροπολογία 17, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 18 και βιομηχανίας 14 υπέρ να τις πάρουμε από κοινού εντάξει 18 και 14 λοιπόν υπέρ κατά εγκρίθηκαν και οι δύο τροπολογία 19 υπέρ κατά εγκρίθηκε βιομηχανίας 15 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 20 υπέρ κατά εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στις ε, ε, σκέψεις. Έχουμε την ε, πρώτη τροπολογία σημαντική για τη συμμετέχει η Επιτροπή Περιφερειών υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 1 τώρα. Κορέιντ Κάμπος υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και έτσι τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά στο το σύνολο του ψηφίσματος ώστε να υπάρχει και επίσημα η καταχώρηση του αποτελέσματος. Η κυρία Ρούλη είναι υπέρ, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον. Σας ευχαριστώ θερμά. Περνάμε τώρα στην έκθεση της πρωτοβουλίας της κυρίας Κόλιν Λάγκεν, που είναι και η παρθενική έκθεση της κυρίας Κόλιν Λάγκεν στην Επιτροπή. Με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας ε, για την καταναλωτική πίστη. Θέλετε, κυρία Συγγετρία, να πείτε κάτι για την έκθεση. Όχι, οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Κύριε Πέντεργας, ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να αποσύρω το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8 που ε, εμένω στο να αντικατασταθεί το sufficient από το important αλλά για το υπόλοιπο τμήμα το δεύτερο θα ήθελα να το αποσύρω. Θα ήθελα να παραμείνει το important, το σημαντικό, να αντικαταστήσει το sufficient, το αρκετό. Με αυτή την αλλαγή είμαι ικανοποιημένη. Το υπόλοιπο τμήμα μπορώ να το υποσύρω από την τροπολογία 8. Ευχαριστώ, Μάλκολμ. Ευχαριστώ. Τροπολογία 7 πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 7. Παρακαλώ, επιταχύνετε λίγο. Εκτός αν έφυγαν ε, αφήνοντας κάρτες τους στα μηχανήματα μερικοί. Παρακαλώ, επισπεύστε λίγο. 13 υπέρ 21 κατά. Απορρίπτεται. Προσοχή στην κυρία Ρούλε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές του κυρίου Μπουσόη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 της ΕΚΟΝ. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα παρακαλώ ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με διαφορά. Δεύτερο τμήμα καλύπτεται από τις μεταγενέστερες παραγράφους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ψηφοφορία κατά τμήματα Τη τροπολογία 8 της κυρίας Πρέντεργκαστ. Τι θα γίνει τελικά. Στο πρώτο τμήμα αντικαθίσταται όρος αρκετός από το σημαντικός. Αποσύρθηκε το δεύτερο τμήμα από την κυρία Πρέντεργκαστ. Καταλάβατε τι ψηφίζουμε όλοι. Ωραία, για το πρώτο τμήμα αντικαθίσταται όρος sufficient από το important. Ποιο είναι υπέρ τη αλλαγή του αρκετός από το σημαντικός. Κατά ε, εμφανώς εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την υπόλοιπη παράγραφα, αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς το δεύτερο τμήμα, δηλαδή. Γιατί το δεύτερο τμήμα το έχει αποσύρει η κυρία Πρέντεργκαστ. Σε ό,τι φορά τις ειδικές πληροφορίες λοιπά Ψηφίζουμε το σύνολο λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της παραγράφου, κατά αποχές εγκρίνεται και εδώ με διαφορά. Τροπολογία είναι της κυρίας Ρούλε με προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία είναι της ΕΚΟΝ καλύπτεται. Τροπολογία 4 της ΕΚΟΝ. Ποιο είναι υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 4 της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Τέλος ψηφοφορίας. 23 ε, κατά, 11 υπέρ απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 έχει αποσυρθεί. Ε, τροπολογία 5, Colin Langen. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 11, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία της ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Με 14 υπέρ, 21 κατά. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 εικόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ, τις 13. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 14 του κύριο Όμπερ Μάιερ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 14 του κυρίου Όμπερμαϊρ. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 21 κατά. Τροπολογία 15, Πρέντεργαστ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά και για την 16 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί δυστυχώ τη τροπολογίε ΕΚΟΝ. Για την τρία τη ΕΚΟΝ άρχεται η ψηφοφορία. Τρίτη τροπολογία τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Τέλος ψηφοφορία. απορρίπτεται. Τροπολογία 6 της ΕΚΟΝ. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6 της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 8 της ΕΚΟΝ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 της κυρίας Πρέντεργα. με προφορική τροπολογία της συγκίτρια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 της κυρίας Πρέντεργα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 της κυρίας Πρέντεργα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 20. Uh, the vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αποχή της κυρίας Ρούλε. Τροπολογία 19. Ψηφίζουμε. 19. Ε, όχι ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 της κυρίας Πρέντεργκαστ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 της κυρίας Πρέντεργαστ. Ηλεκτρονικά για την 22 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 του κυρίου Κάρας. Ποιος είναι υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 23. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. 23. Εκ, τροπολογία Ότμαρ Κάρας. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, ψηφίστε λίγο πιο γρήγορα, γιατί ε, μας έχουν μείνει πολλά ακόμη θέματα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Με την προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 28. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εκόν 11. Ε, ως προστίκη. Ποιος είναι υπέρ. Εκόν 11. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Εκόν 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 της ηγήτριας για τις αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του κ. Σουβάμπ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Αποσύρεται. Τροπολογία 5. Πρέντεργαστ. Με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εκόν α. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται με διαφορά. Εκόν Β υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτό. Εκόν Σ ε, ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Εκόν Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος, του ψηφίσματος μάλλον. Ποιος ε, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, κάποιος έμεινε πίσω. Εντάξει, 33 υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Κυρία Κόνλι Λάγκεν, συγχαρητήρια θερμά, πρώτη σας έκθεση. Μπράβο σας. Περνάμε τώρα... Περνάμε τώρα λοιπόν στην έκθεση την επόμενη για ψηφοφορία του κυρίου Κοφεράτη για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Κύριε Κοφεράτη, θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση πριν την ψηφοφορία, όχι. Συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 47. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά δεκτή. Περνάμε αμέσως στην τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. 50 υπέρ κατά δε, απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 53 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ κατά δεκτή. 55 υπέρ κατά δεκτή. 56 υπέρ Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον ηλεκτρονικά για την 56. Πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ 16 κατά. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Η κυρία Ρόιτεβα. Εγώ ψήφισα κατά, αλλά δεν μπόρεσα να αλλάξω. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα, λέει ο πρόεδρος, δεν μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Παρακαλώ να φροντίζετε έγκαιρα να ψηφίζετε. Συμπιβαστική 9 λοιπόν, υπέρ, κατά, δεκτή. 58 υπέρ κατά δεκτή. 59 υπέρ κατά δεκ, απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά. Τώρα συμβιβαστική 10 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος Δεκτή. 18 υπέρ, 16 κατά. Περνάμε τώρα στην 61. Τέλος. 62 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, δεκτή. 64 υπέρ κατά δεκτή. 65 υπέρ κατά δεκτή. 66 υπέρ κατά δεκτή. 12 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά δεκτή. 14 υπέρ κατά δεκτή. 68 υπέρ κατά δεκτή. 16 συμβιβαστική υπέρ κατά δεκτή. Συνεχίζουμε με την 73 αν δεν κάνω λάθος. 73 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 75 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 17 υπέρ, κατά, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, δεκτή. 78 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, δεκτή. 79 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος. 18 υπέρ 16 κατά γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στην 81. Α, όχι, για μια στιγμή. Έχει καταπέσει 81, οπότε ψηφίζουμε την 20. Την 20 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 82. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Για μια στιγμή ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 82. Πέρα στις ψηφοφορίες. 83 τώρα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 85. Συμβιβαστική 13 ειπε κατά, δεκτή. 2287 από κοινού Είπε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 και 87. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. 88 τώρα υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, δεκτή. 23 υπέρ, κατά, δεκτή. 24 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 24. 25 υπέρ κατά δεκτή. 26 υπέρ κατά δεκτή. 27 υπέρ κατά δεκτή. Η 90 έχει καταπέσει. 91 υπέρ κατά δεκτή. 92 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 94. Άρχεται η ψηφοφορία για την 94. Δεκτή. 95 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά δεκτή. 98 υπέρ κατά δεκτή. 99 υπέρ κατά δεκτή. 100 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά δεκτή. 28 υπέρ κατά δεκτή. 29 υπέρ κατά δεκτή. 30 υπέρ κατά δεκτή. 102 έχει αποσυρθεί, 103 καταπέσει, 31 υπέρ κατά δεκτή. 32. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 32. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά δεκτή. 35 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά δεκτή. 39 υπέρ κατά δεκτή. 40 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά δεκτή. Ε, τροπολογία 1 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική για την τροπολογία υπαρίθμενα. Τέλος της ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά δεκτή. Έχει αποσυρθεί 43, 2 υπέρ καταδεκτή δεκτή. 30. Εδώ γίνεται κατά διέρεση ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. Το σύνολο λοιπόν της νομοδότησης σε ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την γνωμοδότηση Κοφεράτη. 31 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κοφεράτη. Τι μένει τώρα. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γκάλο. Αυτή θα ψηφίσουμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Η κυρία Γκάλο δεν παρίσταται. Περνάμε και ψηφίζουμε άμεσα. Τροπολογία 15 λοιπόν. Φερχάιεν υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 16 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 γκαλό υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 17 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 18 αποσύρθηκε. Η 19 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 20 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 21 αποσύρθηκε. Ο προφορική τροποποίηση στο άρθρο 5 της κυρίας Γκαλό υπέρ κατά εγκρίθηκε. Πού είμαστε τώρα, πού πάμε. Τροπολογία 6 μάλιστα. Τροπολογία 6 Γκαλό υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 25 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 26 υπέρ κατά εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά εγκρίθηκε νομίζω αλλά μια και είναι δική μου τροπολογία θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να μην πούνε ότι ευνοώ την τροπολογία μου άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την δική μου τροπολογία την 27 πέρας ψηφοφορίας τώρα και εγκρίθηκε πράγματι τροπολογία 28 υπέρ. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 28 επίσης. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η τροπολογία 29 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 29. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα και αυτή εγκρίθηκε. Περνάμε και πάμε στην προφορική τροπολογία της κυρίας Τούν και άλλων υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Στα σκεπτικά τροπολογία 1 της κυρίας Γκαλό υπέρ. Κατά Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικά αυτή τη φορά. Τροπολογία 1 της κυρίας Γκαλό. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η ένα. Τροπολογία 7. Φερχέιεν. Να τις πάρουμε όλες από κοινού ομού. Μάλιστα. Εντάξει. Όλες οι τροπολογίες της κυρίας Φερχάγεν έχουν ένα σημείωμα. Τις κύριες κατηγορίες, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ας τα ελέγξουμε. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες 7, 8, την 2, την 9, 11, 12, 13 και 14. Είσαστε ε, σύμφωνοι με αυτό? Όχι. Η ομάδα μου θα ήθελε να ψηφίσουμε κάποιες ξεχωριστά. Ας τις πάρουμε λοιπόν γοργά μία προς μία. Τροπολογία 8, Φερχάγεν, υπέρ, κατά. Ας συγγνώμη. Α, εντάξει, την αγνόησα αυτήν. Ξε, ξαναξεκινάμε. Τροπολογία 7 αυτή τη φορά. Φεχάιεν 7 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 8 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε και αυτή είναι σαφές. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Η τροπολογία 11 αποσύρθηκε. Η 12 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην τελική ψήφιση που άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Και πέρας τώρα της ψηφοφορίας μας η κυρία Ρούλε ψήφισε υπέρ, εν πάση περιπτώσει. 32 λοιπόν υπέρ, το τελικό αποτέλεσμα, καμία αποχή, κα, καμία ψήφος εναντίον, μία αποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια κυρία Γκάλο. Και τώρα περνάμε τέλος στην έκθεση του κυρίου Τσασκόφσκι για την γνωμοδότηση που θα χορηγήσουμε προς την Επιτροπή τη Βιομηχανία την ε, επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 33 καταπίπτει, 34 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 35 Ποιο είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα γιατί έχει αλλάξει ο σχετισμός. Τροπολογία 35 παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 35. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 37 καταπίπτει. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 39. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 17 προς 13 ψήφου. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Σωστά. Ναι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 40 καταπίπτει. Και οι υπόλοιπε μέχρι τη 45. Περνάμε στη 46. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα η 11 καταπίπτει. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία για τα 48. Τέλος. 17 ψήφισαν υπέρ και 14 κατά. Εγκρίνεται. Η 13 αποσύρεται. 49 του είχε το ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51. Η 50 καταπίπτει. Περνάμε στην 51. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 51 μέχρι 55 μαζί. Ωραία. Ποιο είναι υπέρ? 51, 52, 53, 54 και 55. Όχι, δεν συμφωνούνται με την ομάδα ψηφοφορία. Ας τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. 51. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 55 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 56 καταπίπτει. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 16 την αιτιολογική σκέψη 6. Τέλος ψηφοφορίας. 18 ψήφισαν υπέρ και 12 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία για την 17. τέλος. Δεν ψηφίζουν και πολύ όμως. Εγκρίνεται 16 υπέρ. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόεδρε, ξέχασα να ψηφίσω. Είμαι υπέρ. Α, να είστε πιο γρήγοροι. Το σκεφτούμε. Τροπολογία 19, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τώρα παρακαλώ ψηφίστε. Αν ψηφίσετε μετά, είναι αργά. 18 υπέρ, 12 κατά. Τροπολογία 20. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 20 τώρα. Τέλος. 21 υπέρ, 9 κατά. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η αναποσύρεται 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Με διαφορά. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27 κατά πίπη. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28, προσθήκη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει, 29 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά εγκρίνεται και αυτή. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και δύο αποχές. Ευχαριστούμε θερμά τον εισηγητή, τον κύριο Τσασκόφσκι. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Περνάμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Σμιτ. Ε, είστε ευπρόσδεκτοι να παραμείνετε για τη γνωμοδότηση του κυρίου Σμιτ, αλλά αν επιμένετε να φύγετε σώνη και καλά, παρακαλώ ήσυχα. <laughs> Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που είναι το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Όλε Σμιτ, τον οποίο και καλώς ορίζω εγκάρδια, με θέμα τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050. Πριν από καμιά δύο εβδομάδες είχαμε τη συζήτηση, μας υπέβαλε το σχέδιο γνωμοδότησης, θα, ακούσαμε, θα ακούσουμε τον εισηγητή, μετά του και οδησίγητες Μπάστος, Κορέα κάμπο, Ρούλε, Πιέλαν και ένας άλλος Ασκόλικοφ παρόλο που είναι σκιώδη, έφυγε Α το ξαναφέρει κάποιο στην αίθουσα θα συνταχθεί γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Βιομηχανία που αρμόδιος κατ' ουσίαν ε, για την έκθεση είναι ο κύριο Σαβέλα, ο κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπα και στην προηγούμενη μα συζήτηση, το θέμα είναι ζωτική σημασία. Και νομίζω ότι σύσσωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο η Επιτροπή μας ε, καλωσορίζει θερμά τη στρατηγική αυτή, γιατί έχει κεφαλαιόδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις εργασίες. Υπήρξαν κάποια μικροκολλήματα, θα τα θυμάστε όλοι. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει πέντε σενάρια και δέκα συμπεράσματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια αηφόρο ενεργειακή πολιτική τονίζεται ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι μακρόπνοη και μακροπρόθεσμη, ώστε και ο κλάδος και οι πολίτες να ε, έχουν τη βεβαιότητα της προβλεψιμότητας. Και είναι σημαντικό αυτό για τις κρατικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε βιώσιμους τρόπους ενέργειας. Επίσης, σημαντικό είναι να υιοθετήσουμε μια οριζόντια προσέγγιση και ε, σε, όλες τις, ε, σε όλους τους κρίκους αλυσίδας ε, της παραγωγής ενέργειας προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Έχω κάποιες παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, που μπορεί να μην είναι ζωτική σημασία, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικές και καλό θα ήταν να τις συζητήσουμε. Τις επισήμανα και στην πρώτη συζήτηση αφορούν το CCS, δηλαδή το, τη μέθοδο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Η χρήση της μεθόδου αυτής μπορεί φυσικά να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του α, άνθρακα από 85% και πάνω, αλλά δεν επηρεάζει ε, τις... Ε, εκπομπές από τα ορυχεία και αφήνει μάλιστα επικίνδυνα υλικά που θα πρέπει να αποθηκευτούν, όπως συμβαίνει στις, στους πυρηνικούς σταθμούς για παράδειγμα. Οπότε, τι γίνεται με την ενέργεια που απαιτείται για την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Γιατί χρειαζόμαστε όλο και περισσότερα καύσιμα για να παράγουμε το, την ίδια ποσότητα ενέργειας ανάλογα με το είδος του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας. Και Επίσης, έχουμε 24 με 40% περισσότερες ανάγκες ενέργειας, ενώ για τα εργοστάσια φυσικού αερίου είναι 11 με 22% και για τα συστήματα αεροποίησης που χρησιμοποιούν άνθρακα είναι 14 με 25% οι πλέον ανάγκη ενέργειας. Βέβαια, έχουμε και τα περιβαλλοντικά προβλήματα εξαιτία ε, της εξόριξης ε, άνθρακα και φυσικού αερίου. Στη διάσκεψη των κλιματικών αλλαγών το 2011 στο Τέρμπαν ε, των Ηνωμένων Εθνών καταλήξαμε σε συμφωνία να υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά αυτά τα σχέδια με το μηχανισμό CDM, ε, το μηχανισμό δηλαδή της καθαρής ανάπτυξης. Βέβαια το κόστος παραμένει αβέβαιο και μάλιστα ε, αναμένεται δραστική αύξηση των τιμών εξαιτής τη χρήση τη και αποθήκευση του άνθρακα. Επίσης, αν προσθέσουμε και το κόστος των επενδύσεων αλλά και την περαιτέρω χρήση ενέργειας, ε, οδηγούμαστε σε ένα υπέραγο κόστος για το CCS. Χρειαζόμαστε περισσότερα καύσιμα, υπάρχει το κόστος αποθήκευσης, οπότε ε, θα αυξηθεί και η τιμή της ενέργειας που παράγεται. Και το συμπέρασμά μου ή το ερωτηματικό που θέτω είναι ότι θα έπρεπε πιστεύω να εξετάσουμε τα αποτελέσματα αυτά με ιδιαίτερη προσοχή προτού καταλήξουμε σε αυτή την κατεύθυνση και πορευτούμε αυτή την πορεία. Μετά έχουμε γενικότερα τα θέματα του κόστους επίγουσα δράση μπορεί να διασφαλίσει ότι τα υψηλότερα κόστη στη συνέχεια θα μπορέσουν να αποφευχθούν. Συμφωνώ με αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κόστος θα αυξηθεί όσο περισσότερο περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια και επ' αυτού είναι σαφή η Επιτροπή. Δεν προσπαθεί να αποκρύψει αυτό το πρόβλημα καθόλου οι μείζονες επενδύσεις που θα οδηγούσαν σε αυξημένο κόστος ούτως ή άλλως πρέπει να γίνουν διότι έχουμε εδώ υπερήλικες ε, υποδομές ε, και μονάδες παραγωγών και αυτό δίνει την εξαιρετική ευκαιρία να γίνουν οι βέλτιστες επιλογές αυτό τονίστηκε αυτό από την Επιτροπή την τελευταία φορά συμφωνώ απόλυτα η αποδοτικότητα ενέργειας είναι ένα ε, υψηλά αποτελεσματικό μέτρο για να καταφέρουμε αυτό το στόχο και θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην όλη συνολική αλυσίδα της, ε, του εφοδιασμού με ενεργειακά προϊόντα. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια χαμηλού επίπεδου οικονομία άνθρακα ε, ως ευκαιρία αυτό για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκόσμια. Η εσωτερική αγορά τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον πρωτοπόρο ρόλο της σε σχέση, συγγνώμη, τον ρόλο πρωτοπόρου που έχει για να καταδειχθεί πώς μπορεί μια φιλόδοξη πολιτική για την προστασία του κλίματος μπορεί να συνδυαστεί με οικονομική ανάπτυξη. Και νομίζω έχουμε αρκετά καλά θετικά παραδείγματα εδώ ενώπιον μας, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες μας θα έλεγα. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να υλοποιηθούν τα ήδη ενισχύει νομοθετικά μέτρα και σε σχέση και με το πρόσφατο πακέτο για την ενεργειακή αγορά πρέπει μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά να επιτευχθεί από πλευράς Ευρώπης. Ε, φυστάται η προσοχή ότι η καταληκτική προθεσμία είναι ήδη το 2014. Πρέπει να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να εργαστούμε έντονα για να τα καταφέρουμε μέχρι τότε. Ε, αυτή πρέπει να είναι λοιπόν η πορεία μας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην Ευρωβουλή γενικότερα. Αυτό το μέσο θα πρέπει να συμπληρώνεται με τις αναγκαίες δράσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη π.χ. στρατηγική για τον ορίζοντα 2020. Μείωση των εκπομπών ρήπων του ε, θερμοκηπίου ώστε να να καταλήξουμε σε μια πιο αποτελεσματική αγορά. Είναι μια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που εργάζονται ή ενδιαφέρονται για την αγορά ανανεώσιμων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στους καταναλωτές. Και εδώ φυσικά θα έλεγα αυτή είναι η κυρία επικέντρωση, η κυριότερη εστίαση ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή για μας σε αυτό το θέμα στους καταναλωτές για το πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τις συνήθειες στην κατανάλωση ενέργειας. Στη χώρα μου παράδειγμα σήμερα μας λένε και μαθαίνουμε τη λάντσα και το πλήσιμο των ε, πιατικών να την κάνουμε το βράδυ. Θέματα όπως τέλει για τον άνθρακα και τις εκπομπές άνθρακα έχουν σημασία σοβαρή, ως το τέλος, τέλος όμως θα επιβαρύνουν τους πολίτες ως προς αυτά νομίζω ότι μπορούμε να αυξήσουμε αυτά τα τέλη, γιατί είναι ένα καλό μέσο αυτό, εν πάση περιπτώσει, για μας ως καταναλωτές να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα τελικά κόστη και να αντιμετωπιστούν αυτά λύσεις όπως ευφυή δίκτυα σε αυτή την ε, ανακοίνωση για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ε, και σε σχέση με τους παρόχους ε, μπορούν οι καταναλωτές να παρατηρούν το κόστος και να μπορούν έτσι να υποφεληθούν. Και δίνω και κάποια παραδείγματα σχετικά. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μεσοπρόθεσμη διαμόρφωση των τιμών θα αυξηθούν οι τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα, άσχετα ποια πολιτική θα συμφωνήσουμε εμείς. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ αυτών που γίνονται για την ενεργειακή πολιτική και αυτών για την κοινωνική πολιτική και αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι τα θέματα της φτώχειας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και όχι με την ρύθμιση των τιμών ενέργειας. Καλύτερα μπορούν να στοχοθετηθούν αυτά τα θέματα σε επίπεδο κρατών μελών. Τουλάχιστον αυτή είναι η πείρα που συνέλεξα εγώ, αυτό είναι το βίωμά μου ως ενεργού πολιτικού στην ίδια μου τη χώρα, σε όλα τα επίπεδα, σε 35 ολόκληρα χρόνια υπηρεσίας του στο λειτουργήμά μου. Αυτά είναι και ολοκλήρωσα, Πρόεδρε. Και καταλήγω τώρα στο πιο ευαίσθητο ζήτημα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συνένεση σε αυτά τα θέματα επί σχεδόν όλων των θεμάτων. Όμως εδώ είναι το ένα θέμα που πιστεύω ότι ούτε θα μπορούσαμε ούτε θα έπρεπε και να συμφωνήσουμε επ' αυτού, διότι έχουμε διαφορετικές απόψεις ούτως ή άλλως γι' αυτό. Και αυτό αφορά φυσικά την πυρηνική ενέργεια. 30 χιλιόμετρα, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων ζω από ένα πυρηνικό αντιδραστήρα και οι Δανείοι τον έκλεισαν και στη χώρα μου έστω κιόλας διότι από την πρωτεύουσα, από την Κοπενχάγη το αντιμετώπισαν το θέμα αυτό και κανένας δεν βρέθηκε που να πει ότι αυτοί δεν είναι οι λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να κλείσει ο ποινικός αντιδραστήρας. Το να ζητηθεί τώρα από μια άλλη χώρα όπως έγινε να γίνει αυτό ε, και υπήρξε μια συναλλαγή. Ε, να πήραμε τη γέφυρα που μας έδωσαν Γερμανοί προς ε, Δανία. Διαφορετικά δεν θα γινόταν αυτή η γέφυρα. Και έτσι έκλεισε αυτός ο ποινικό αντιδραστήρας. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω φυσικά ότι θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να καταφέρουμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας. Φυσικά όμως από την άλλη πλευρά να απαιτήσουμε το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Όμως είναι μια αυταπάτη θα έλεγα να λέει και να πιστεύει κανείς ότι και αυτό τουλάχιστον όχι για τα επόμενα 50, 60, 70, ίσως επόμενα 100 χρόνια ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη. Λοιπόν, στη Γερμανία κυρία Αρβίλα, έστω, το κάνατε εσείς αυτό και είπατε θα κλείσετε τους πυρηνικούς σας αντιδραστήρες. Και αυτό τι κάνει, αφήνει περισσότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα για τους υπόλοιπους, για μας, για τον Βορρά και Τώρα, για την χρήση μεγαλύτερη ποσότητα ρωσικού φυσικού αερίου κτλ. Η Γερμανία και η Ιαπωνία είναι οι μόνε που πήραν την απόφαση να κλείσουν του πυρηνικού αντιδραστήρε. 435 έχουμε πυρηνικού αντιδραστήρε συνολικά παγκόσμια. 65 βρίσκονται υποκατασκευή. Και έχουμε μεταξύ άλλων και στην Φινλανδία αυτό το φαινόμενο. Και πολλές χώρες ε, χτίζουν, δημιουργούν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Θα ήθελα να πω όλων τούτων λεχθέντων ότι μπορεί κανείς να είναι πολύ φιλοπεριβαλλοντικός και βιώσιμος στην αηφορία του λέγοντας ότι αν είχαμε μια νέα γενναία πυρηνικών αντιδραστήρων που θα λειτουργούσαν, αυτό θα ήταν ένα θεμελιώδες στοιχείο για να αντιμετωπιστούν βιώσιμα οι περιβαλλοντικές αλλαγές στην Ευρώπη και παγκόσμια. γνωρίζω τα επιχειρήματα και τα σέβομαι βέβαια, αλλά θα ολοκλήρωνα επ' αυτού λέγοντας, Πρόεδρε, ότι πιστεύω ότι η απόφαση που ελήφθη από τη Γερμανία δείχνει την έλλειψη, έλλειψη, απουσία επίπεδου λήψης απόφασης στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω ακόμα και αν ο Επίτροπος, παρότι ο ίδιος είναι Γερμανός, αν γνώριζε το τι συνέβαινε. Είναι θλιβερό αυτό. Και ο κύριος Χατζημαρκάκης απουσιάζει τώρα βέβαια Νομίζω αυτό δείχνει ότι και η φιλελεύθερη ομάδα στη Γερμανία, το κόμμα των φιλελευθέρων, το δέχτηκε αυτό. Γιατί έγινε αυτό εν εθρία και κανείς δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και εμείς οι γειτονικέ χώρες τι θα κάνουμε, θα πρέπει να υπομισθούμε αυτό το πρόβλημα, να ζήσουμε με αυτό, όπως φυσικά και οι Γερμανοί. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Δεν θα καταλήξουμε σε συνένεση σε αυτό το σημείο. Ελπίζω όμως ότι μπορείτε να σεβαστείτε την δική μου προσέγγιση και τι ιδέε μου. Και εγώ οπωσδήποτε θα σεβαστώ τι δικέ σα Ευχαριστώ. Uh, Πράγματι, πρόκειται για μια ευρυτάτη παρουσίαση. Είναι μεγάλη χαρά που σας είχαμε σαν εισηγητή, γιατί έτσι έχουμε τώρα κάπως ξεκάθαρες ιδέες για το τι θα συζητήσουμε θα έπρεπε να καλωσορίσω τον κύριο Βένστροπ από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, θα του δώσω το λόγο αργότερα. Ας ξεκινήσουμε όμως με τους Σκιώδης και με την κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την ε, πολύ σαφή παρουσίαση που μας έκανε της ε, πολύ τεκμηριωμένης έκθεση, ε, μα μίλησε για, την, ε, ε, για τον ανεφοδιασμό σε άρθρακα, για την, για την οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα, για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, για του καταναλωτέ, για το σύστημα δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και το καθεξή. τώρα, θα ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο, το θέμα τη πυρηνική ενέργεια. Στην τελευταία ανταλλαγή απόψε στην Επιτροπή μα. ακούσαμε ξεκάθαρα από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 2005, μάλιστα η πυρηνική ενέργεια ε, θα ε, λάμβανε ε, πολύ μικρό ρόλο, περιφερειακό ουσιαστικά στην παραγωγή ενέργειας. Είχαμε όμως μία τριανταεκοδετία για να εξετάσω αυτό το θέμα. Δεν έχουμε εστιαστεί αρκετά στο θέμα τη σημασία τη πυρηνική ενέργεια και μάλιστα υπό το πρίσμα και του καταναλωτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει στη γνωμοδότησή μα να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και να μην μιλήσουμε τόσο εκτεταμένα για την πυρηνική ενέργεια. Χαίρομαι για την αναφορά που έγινε των smart grids, των ε, εφιών δικτύων που θα ωφελήσουν τους καταναλωτές αλλά και χαίρομαι που αναφέρεται ως υποχρέωση ε, των ε, παρόχων. Η χρήση αυτών των δικτύων θα μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές. Μην ξεχνάτε ότι εκπονούμε μια γνωμοδότηση που θα συμπεριληφθεί σε μια ευρύτερη έκθεση θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τις δικές μας προτεραιότητες. Μας ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή, το συμφέρον του καταναλωτή και πολύ σωστά συνέταξε την παράγραφο 3 ο εισηγητής στο σχέδιο γνωμοδότης. Ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τώρα και στο μέλλον θα διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην εσωτερική αγορά. Και χαίρομαι που η γνωμοδότηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε κάπως πιο ε, σαφής ε, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική μέσω της ενεργειακής πολιτικής. Το σημείο 9 της γνωμοδότησής σας ε, ίσως θα πρέπει να διατυπωθεί Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιες είναι οι σκέψεις για το σημείο 9, πώς θα μπορούσαμε ίσως μέσω κάποιας τροπολογίας να αναδιατυπώσουμε το σημείο 9. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της διαπαιδαγώγησης ε, των καταναλωτών και της σωστής ενημέρωσης ε, για τους καταναλωτές. Γιατί στο μέλλον η σωστή ενημέρωση θα αποτελέσει ε, ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής. Και είναι προφανές ότι με καλύτερη ενεργειακή πολιτική θα αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά είναι ίσονο σημασίας. Αφορούν, επαναλαμβάνω, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, το μέλλον της ε, ε, μέσο και, και μακροπρόθεσμα και το θέμα της ενημέρωσης ε, και διαπαιδαγώγηση κατά κάποιο τρόπο ε, των καταναλωτών. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε εύκολα συμφωνία με τον εισηγητή για τα θέματα αυτά. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Κορέα Ντεκάμπος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο Όλε Σμιτ για το καταπληκτικό του έργο, αλλά να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιόλογη της πρόταση στρατηγικής για τον ενεργειακό τομέα. Όπως είπε ο κύριο Σμιτ, έχουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας, γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε κοινούς κανόνες και διατάξεις που θα είναι διαφανείς, ανταγωνιστικές, και εναρμονισμένε. θα ακολουθούνται από όλε τι χώρε. και μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε του στόχου τη βιωσιμότητα, τη χρησιμοποίηση των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τη συνεργασία των εθνικών αρχών εποπτεία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικέ τιμέ για τον καταναλωτή. Ε, ακόμη και αν είχα αμφιβολίες για την αρχή αυτή, ε, διασκεδάστηκαν τι τελευταίε πέντε μέρε που ήμουν στην Ιαπωνία και που συμμετείχα σε έντονες συζητήσεις για τα θέματα της ενεργειακής πολιτικής και την πραγματική ε, απώλεια ανταγωνιστικότητας, την ε, απώλεια της διαφάνειας και την επικάλυψη, κάτι που οδήγησαν σε έλλειψη ε, σωστής κρίσης, κάτι που οδήγησε στο, στη δεύτερη καταστροφή της Φουκουσίμα, μετά το παλιρακό κύμα. Το θέμα της διαφάνειας στην αγορά είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί η αγορά να μην είναι υπανάκια, αλλά είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός προειδοποίησης, συναγερμός για το πρόβλημα αυτό. Δυστυχώς δεν ε, λειτουργήσε το σύστημα αυτό στην Ιαπωνία εξαιτίας καρτελοποίησης του συστήματος. Σημαντικό και το θέμα του ενεργειακού μείγματος. Παρόλο που αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, θα πρέπει να γίνεται με βάση κοινού στόχους και μια συντονισμένη ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε τους ε, στόχους μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη και το τελικό αποτέλεσμα που είναι εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Το είναι και το αντικείμενο της δικής μας επιτροπής, η μέρημνα για τον καταναλωτή και σε όλες τις γραμματοτήσεις μας θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Επίσης, να εστιάσουμε την προσοχή της Ένωσης και των κρατών μελών σε ε, επενδύσεις υποδομές που θα εξασφαλίζουν ε, προστασία και ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού και θα Δίνουμε έμφαση τέτοιου μακροπρόθεσμε επενδύσει, συνδυασμό με συγκεκριμένα κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα και κατάλληλε ιστορικέ πολιτικέ. Έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο ενεργειακής αλληλεπίδρασης. Είναι σημαντική αυτή η μέρημνα για να αντισταθούμε στην, στον πειρασμό των κρατών μελών να, να επανεθνικοποιήσουν αυτό το θέμα και να ε, κλείνουν τις αγορές τους. Είναι σημαντικό επίσης ε, να οδηγηθούμε σε μια αποσυμφόρηση των υποδομών, να άρουμε τις στενοπούς και να, να οδηγηθούμε σε μια πραγματική ενεργειακή ολοκλήρωση, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές σχέσεις. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ε, διατάξεις που θα διευκολύνουν τις νέες εισόδους στην αγορά. Μην ξεχνάτε ότι οι πολιτικές της, ε, και οι αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος. Γι' αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή στα δίκτυα. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διακοιμάνσεις ε, στις χρήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ Βορρά και Νότου. Και μόνο μια ε, συμμετοχή και ολοκλήρωση των δικτύων μπορούμε να οδηγηθούμε σε καλύτερη αποθήκευση και σε μια πιο αδιάλειπτη μεταφορά ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την τον παραβαλλοντικό αντίκτυπο του στήματο δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, εξακολουθούν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την τεχνολογία αυτή. Έχουμε και άλλε προτάσει για το μη συμβατικό ή το σχιστολιθικό αέριο. Θα είναι σημαντικό για να μειωθεί η εξάρτησή μα από άλλε χώρε και ιδιαίτερα τη ΣΥΠΑ σε ορυκτά καύσιμα. Βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε σχολαστικά τη χρήση της τεχνολογίας χιστολιθικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπό το φως και του πιθανού αρνητικού περιβαλλοντικού αντικτύπου. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένα θέμα που μας βρίσκει όλους σύμφωνους και επηρεάζει άμεσα και την ε, άνεση των καταναλωτών. Είναι σημαντικό επίσης ε, να προσέξουμε τι θα γίνει με την ε, σταδιακή μείωση του άνθρακα μέχρι το 2050. Οι ενεργειακές και ε, δαπάνες και δαπάνες των μεταφορών θα αποτελούν και μεγαλύτερο τμήμα του, προπολογισμού και των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Υπάρχει μια οδηγική πορεία και θα πρέπει να την ε, μετριάσουμε χάρη σε κατάλληλη ρύθμιση των κρατικών νομοθεσιών και μια προσπάθεια στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, άσχετα με τις προσωπικές απόψεις του καθενό, άσχετα αν ήταν καλή κακή η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρηθεί η πυρηνική ενέργεια είναι θέμα επικουρικότητας. Είναι προφανές ότι δεν είναι θέμα επικουρικότητα η πυρηνική ενέργεια, αλλά απόλυτης ολοκλήρωση. Εν πάση περιπτώσει, άσχετα με την απόφαση που ελήφθη για το θέμα αυτό, πιστεύω ότι ο πυρηνική το θέμα της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας είναι στο μέσο το οποίο δεν θα πρέπει να αποποιηθεί των ευθυνών της ή να παραιτηθεί της αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα των ελέγχων αντοχής και ε, ελέγχου σε περίπτωση ακραίων συνθηκών για τα πυρηνικά εργοστάσια είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο εκεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Θέλω ρητά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όχι μόνο για την εξαιρετική έκθεση, αλλά επίσης και για αυτό που εδώ προτείνει, αυτά που προσωπικά ανέφερε ο ίδιος. Θέλω για άλλη μια φορά ρητά και κατηγορηματικά να τονίσω κύριε Σμιτ ότι στην κριτική σας, στην απουσιάζουσα, ελίπουσα στρατηγική στο ευρωπαϊκό επίπεδο συμφωνώ απόλυτα. Και θα συμφωνούσα και μαζί σας αν, αν λέγατε και όταν λέτε ούτε η Γερμανία έχει αυτή τη στρατηγική που είναι αναγκαία και θα ήταν αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε την ε, όλο και πιο προχωρημένη, τις ε, όλο και πιο προχωρημένες αλλαγές ε, του κλίματος. Χρειάζεται λοιπόν κατεπηγόντως αυτή η στρατηγική. Ακριβώς σε μια περίοδο που έχουμε μια χρηματοοικονομική κρίση και έχουμε περιορισμό κονδυλίων, πολύ μεγάλη σπανίδα κονδυλίων, να δούμε πώς θα επενδύσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για την ασφάλεια του εφοδιασμού μας σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα και τα δίκτυα, αλλά προς όφελος των καταναλωτών κυρίως. Σε όλα αυτά τα σημεία συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στον τομέα ίσως και πιο πριν κάτι άλλο. Συμφωνώ ρητά μαζί σας επίσης και στις επικρίσεις που διατυπώνεται στο σημείο 5 όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα. Και εδώ πιστεύω ότι κάπως ένα πείραμα καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να έχει σκεφτεί ποια είναι τα κόστη, ποιε είναι οι επιπτώσεις, ποια είναι τα κονδύλια τα οποία δεν θα μπορέσουν διαφορετικά να χρησιμοποιηθούν αν τύχουν αυτή τη χρήση. Όταν πιεζόμαστε σε σχέση με τα κονδύλια πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά σε σχέση με τα χρήματα που σπανίζουν. Για τα πυρηνικά εργοστάσια, του πυρηνικού αντιδραστήρε έχω μια διαφορετική θέση και θέλω να το πω ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια διαφανή αγορά θα πρέπει φυσικά και στην ατομική πυρηνική ενέργεια να συμπεριλάβουμε όλα τα αναγκαία κόστη ασφάλισης και ασφαλίσεων για να ε, αντιμετωπιστούν πιθανότητες ε, που μπορεί να ε, μην πάνε καλά στο μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό για να υπάρχουν αποθέματα ασφάλειας ε, που δεν μπορούν ε, οι καταναλωτές να κληθούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες αν κάτι πάει στραβά. Αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Και το θέμα της αποθήκευσης των αποβλήτων. Και βλέπουμε εδώ και το θέμα με τις δοκιμές stress tests που έγιναν. Δηλαδή αν ε, ερχόταν αυτή η κατάσταση τότε θα ήταν πολύ ακριβότερα τα κόστη. Αυτό είναι το, η μία μου παρατήρηση. Η δεύτερη, εκεί που πρέπει να υπάρξουν κάποιες συμπληρώσεις, θα έλεγα το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα πρέπει κάπως περισσότερο να τονιστεί. Αλλά εκείνο που είναι πιο σημαντικό για μένα, προέρχομαι από τη Βάδη Βιρτεμβέργη, από αυτό το κρατήδιο. Πηγαίνοντας από εκεί προς το Στρασβούργο, βλέπει κανείς ε, τις νέες προκλήσεις. Παντού έχουμε φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες των σπιτιών μας. Η αποκέντρωση δηλαδή σε του ενεργειακού ανεφοδιασμού έχει προχωρήσει πολύ στην ε, Βαδιβιρτεμβέργη. Απ' την άλλη πλευρά είμαστε ένα υψηλά βιομηχανικό, βιομηχανοποιημένο κράτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά, όχι μόνο στα δίκτυα, αλλά και στη δυνατότητα αποθήκευσης, διότι η ηλιακή ενέργεια οδηγεί στο κάποιοι ε, ε, κάποιες μονάδες ε, πετρελαίου για παράδειγμα ή άλλες δεν αξίζουν πια χρηματοοικονομικά. Οικονομικά δεν μπορούν να είναι κερδοφόρα διότι μέσω της έντονης χρήσης της ηλιακής ενέργειας δεν μπορούν να καλύψουν τα κόστη τους. Λοιπόν υπάρχουν νέες, τεράστιες νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να δούμε πώς θα πορευτούμε την αποκεντρωμένη πορεία π.χ. στα φωτοβολταϊκά με την ασφάλεια τον ανεφοδιασμό και με τις επενδύσεις για την αποθήκευση. Αυτά όλα είναι πολύ πιο σημαντικά θέματα, τα οποία θα έπρεπε πιστεύω να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντί του θέματος της σύλληψης και αποθήκευσης άνθρακα, χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης ε, και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που σε όλες τις ώρες της ημέρας ε, του 24ου θα διασφάλιζε την ε, ενέργεια που χρειαζόμαστε και όχι μόνο όταν θα λάμπει ο ήλιος. Χρειαζόμαστε και σε άλλους τομείς. Και στη Βάδη Βιρτεμβέργη έχουμε ενδιαφέροντα ε, θέματα ε, και έχουν υπάρξει σημαντικότερες επενδύσεις στη Βάδη ε, Βιρτεμβέργη για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις χαμηλότερες εκπομπές ρήπων. Λοιπόν. Όλα αυτά την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά την καθορίζουν με καθοριστικό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα πράγμα θέλω να πω γιατί πάντα αναφέρεται ότι σε εμά ή ότι εμείς πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί, διότι προάγοντας την αηφορία στα ενεργειακά θέματα, σε πρώτη γραμμή η θέση των ε, ηλιακών αυτών πάνε στην Κίνα, λέει, προάγεται. Αν δει κανεί τα πράγματα, πρέπει να διαπιστώσει τουλάχιστον 50% της πρόσθετης ε, ενέργειας που παράγεται, παράγεται σε σχέση με τους χειρόνακτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στη χώρα μας, με την εγκατάσταση τέτοιων ηλιακών πάνελ. Και όταν τα δει κανείς, τα υπόλοιπα 50% από τα υπόλοιπα 50% πάλι 30% καταλήγουν στην Ευρώπη διότι οι Κινέζοι αυτά τα πάνε τα παράγουν με μηχανές ε, με βοήθεια μηχανών που παράγονται στην Ευρώπη αυτές οι μηχανές, αυτός ο εξοπλισμός. Και πάλι λοιπόν εδώ να είμαστε διαφοροποιημένοι, να διαφοροποιούμε τα πράγματα σε σχέση με τα πάνελ που ε, ασκούνται επικρίσεις έναντι των Κινέζων. Εντάξει, να είναι φθηνότερα και όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούνται, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση ότι η παραγωγή αξίας παράγεται σε διαφορετικά επίπεδα και όχι μόνο με την άμεση αγορά αυτών των πάνελ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετό χώρο σήμερα για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπίλαν είναι ο τελευταίος ομιλητής ε, για το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, σχεδόν έχουμε εξαντλήσει ε, το χρόνο που προβλέψαμε για αυτή τη συζήτηση. Θα είμαι λακωνικός. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το πολύ μεστό σχέδιο γνωμοδότησης, πολύ ισορροπημένο και τον ευχαριστώ για τα σημεία που συνέταξε και ε, συμφωνώ και εγώ με το σημείο 3, το χρειαζόμαστε ε, ανοιχτή, διαφανή, ενοποιημένη και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας. Και χαίρομαι και για το σημείο 6 που μιλάει για το ρόλο των εφιών δικτύων, των smart grids. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας, γι' αυτό και συμφωνώ και με την παράγραφο 7. Ε, παρόλο που είμαι Πολωνός και η Πολωνία ε, άσκησε βέτο για το έγγραφο αυτό, χαίρομαι και για την παράγραφο 8 του σχεδίου γνωμοδότησης, γιατί ε, λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα των χωρών ε, για τις οποίες ε, ο ρόλος του άνθρακα είναι πολύ σημαντικός. Η κυρία Ρούλε μίλησε για τον ρόλο από μη συμβατικές πηγές ενέργειας και πιστεύω θα πρέπει να το συνδυάσουμε με το σημείο που αφορά το ρόλο των ευφυών δικτύων αλλά και το θέμα της λήψης υπόψης προσ Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορεί να υποβάλλω δύο-τρει τροπολογίε, αλλά γενικώ συμφωνώ με το έγγραφο γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους και Ο κύριος Σβάπ ζήτησε τον λόγο. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλο να λάβει τον λόγο στη συζήτηση. Ο κύριο Σβάπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαρίστω θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό το οποίο είπε ο Λεσμίτ σε ένα σημείο, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, λέει, συμφωνία. Και βρίσκω και σε πολλέ διεξοδικέ ε, και περίπλοκε ε, διατυπώσεις υπάρχει μία σε βάθο ε, αιτία που έχει παραμείνει στο περιθώριο. Ακόμα και αν στο ένα σημείο στο τέλο δεν καταλήγει επί τη ουσία σε, μία, σε καθορισμό μια θέση, πρέπει να είναι σαφέ όμω ότι οι κίνδυνοι στην Ευρώπη σήμερα είναι παντού οι ίδιοι, διότι του πυρηνικού αντιδραστήρε δεν μπορεί να τους σβήσει σε μια χώρα Παγκόσμια υφίστανται αυτοί οι κίνδυνοι όπου λειτουργούν τέτοιοι αντιδραστήρε. Γι' αυτό ξεχωριστή εθνική πορεία και στην ενεργειακή πολιτική αλλά και στου πυρηνικού αντιδραστήρε δεν είναι μακροπρόθεσμη ούτε ε, ασφαλή προοπτική μακροπρόθεσμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε την ενεργειακή εσωτερική αγορά που πρέπει να επιτευχθεί και το, αυτό που αναφέρθηκε για τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην άλλη πλευρά της Βαλτικής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως διασυνοριακό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έτσι αυτό και ε, για τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Κάποιες άλλες χώρες δεν ε, το σκέφτηκαν αυτό και δεν αντέδρασαν ε, σωστά. Και υφίστανται αυτοί οι αντιδραστήρες και ο κίνδυνος και μέχρι τη μελέτη του κυρίου Έτιγκερ δεν έχει καθόλου μειωθεί αυτός ο κίνδυνος και πρέπει να επενδύσουμε στην ασφάλεια. Στο τέλος τέλος όμως δεν θα επιτευχθεί εκείνο το επίπεδο ασφάλειας που άλλοι επιτυγχάνουν. Και γι' αυτό εν πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια κοντόφερη πολιτική μπροστά μας. Και αν θέλει κάποιος με την έκθεση του κυρίου Σμιτ κάτι να αλλάξει, τότε εγώ ως ε, ε, μέλος της ομάδας του ΕΛΚ και το είπε η κυρία Μπάσος, είμαι πρόθυμος να συνεισφέρω. Ευχαριστώ. Ε, Δύο επιπλέον σχόλια. Είναι ενδιαφέρον το έγγραφο της Επιτροπής και ανάλογα με τις απόψεις που έχει κανείς βέβαια Πρέπει να πούμε ότι διευκρινίζει το έγγραφο ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μια σημαντική πηγή και θα είναι μια σημαντική πηγή και το 2050 για την παραγωγή ενέργειας και θα είναι τμήμα πάντα του λεγόμενου energy mix. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας σε αυτό το μείγμα μορφών παραγωγής και τίθεται βέβαια και το θέμα ε, της ε, συγκέντρωσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα και της αποθήκευσής του. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστές είμαστε σε σχέση με όλα αυτά. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο βασικά σκέλη τη στρατηγική μας και αν δεν καταδικάσουμε το σύνολο της στρατηγικής, που δεν το θέλουμε βέβαια, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε σχέση με τις λύσεις που έχουμε μπροστά μας. Να σχολιάσω επίσης ότι μία από τις βασικές δράσεις στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς είναι να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά για την ενέργεια. Αυτό πλέον θα πρέπει να είναι ένας βασικός πολιτικός στόχος και είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να το πετύχουμε έτσι ώστε να λειτουργήσουν με επιτυχία όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η εσωτερική αγορά και να δώσουμε και τα σωστά κίνητρα βέβαια για την στρατηγική. Το ότι δυσκολευόμαστε τώρα δεν είναι καλό μήνυμα θα έλεγα. Είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα. έχουμε κάποιο χρόνο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουμε την άποψή της. Ο κύριος Βέστροπ θα ήθελε να σχολιάσει αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Κάτι το οποίο ακούστηκε από πολλά μέλη είναι η σημασία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Με αυτό φυσικά θα συμφωνήσουμε. Το περιλαμβάνουμε και στη δική μας ανακοίνωση. Η μεταβατική περίοδος θα είναι πολύ περίπλοκη αν δεν λειτουργεί πλήρως η εσωτερική αγορά για την ενέργεια. Εμείς θα υιοθετήσουμε την ανακοίνωσή μας για την αγορά ενέργειας τον επόμενο μήνα θα έχουμε τις τελικές προτάσεις μέχρι το 2014. Νομίζω ότι η ανακοίνωσή μας θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και θα συνεισφέρει και θα συμπληρώσει την έκθεση του Κοινοβουλίου. Σχετικά με το κόστος τώρα και τις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας από τις διαδικασίες αυτές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, το αντιμετωπίζουμε με σοβαρό νομίζω τρόπο θα, υπάρξουν αύξηση, θα υπάρξει αύξηση του κόστους έτσι και αλλιώ λόγω της ανάγκης αντικατάστασης α, κάποιων μονάδων και κάποιων υποδομών που βρίσκονται πλέον σε φάση γύρανσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στην τιμολόγηση της ενέργειας και για τα νοικοκυριά αλλά και για τη βιομηχανία για το CCS τώρα και για την πυρηνική ενέργεια. Το CCS όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από τα τεχνολογικά και το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν με αυτού του τύπου τη τεχνολογία. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε εδώ ότι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτές τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει στο NER 300 θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού και θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την ευθύνη συγχρηματοδότησης. Για την πυρηνική ενέργεια ήταν θετική η διευκρίνηση που έκανε ο Πρόεδρος στο τέλος της ανταλλαγής απόψεων. Εμείς δεν είπαμε ότι η πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει και θα είναι μία αναπλήρωση ενέργεια για το 2050. Υπάρχουν πολλά σενάρια, θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις, τις πολιτικές τις οποίες θα πάρουν τα κράτη-μέλη και όπως είπε ο Πρόεδρος, η πυρηνική ενέργεια θα παίξει ρόλο σημαντικό στις χώρες όπου θεωρείται αποδεκτή τεχνολογία. Η ασφάλεια φυσικά των πυρηνικών εγκατεστάσεων και γι' αυτό εδώ και δύο εβδομάδες δημοσιεύσαμε τα λεγόμενα τεστ αντοχής. Θα γίνουν και νέες πρωτοβουλίες τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται στον τομέα να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται όντας συμβατά πάντα με αυτά τα οποία η ζήτηση καθορίζει. Θα περιμένετε νομίζω την ανακοίνωσή μας πριν από την ψηφοφορία στην οποία θα περάσετε. Λοιπόν κύριε Σμιτ θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση και να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα για την ομοδότησή σας. Όλε Σμιτ. Δεν μπορώ να παρουσιάσω μια περίληψη αυτών που άκουσα, δεν είμαι αρκετά έξυπνος, λέει ο κύριος Σμιτ. Να πω όμως ότι αναφέρομαι πάντα στα θέματα της πυρηνικής ενέργειας γιατί είμαι πολιτικός και γνωρίζω ότι είναι κεντρικό θέμα, πολιτικό θέμα Μπορεί να πείτε ότι τα, τα διαβάσατε αυτά τα οποία σας προτείνω, τα εξετάσατε, αλλά παρόλα αυτά το θέμα είναι όχι τεχνικό, πολιτικό. Σε όλες τις εκλογές, είτε πολιτικές είναι, είτε, είτε βουλευτικές, είτε ε, τοπικές, το θέμα θα, θα έρχεται πάντα στην επιφάνεια. Και στις ε, περιφερειακές εκλογές στην Γερμανία, και στην Βάδη Βιτερβέργη, στις εκλογές που έγιναν ε, τέθηκε το θέμα της Atomkraft, λέει στα γερμανικά, της πυρηνικής ενέργειας. Λοιπόν, όλα επηρεάζονται από αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ψευδέστηση και αυτή είναι η άποψή μου, γιατί έχουμε προβλήματα και στη δική μου χώρα. Η Greenpeace χθε, σαν παράδειγμα, μπήκε σε δύο μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και δεν τους, ε, δεν τους συνέλαβε κανείς. Ε, καταστροφική ασφάλεια στη δική μου χώρα των πυρηνικών μονάδων. Δεν μπήκαν βέβαια στον πυρήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν είναι όλοι ε, τόσο πεισμένοι όσο εγώ γύρω από το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Θα δούμε λοιπόν. Ένα άλλο θέμα είναι το κόστος. Τα κόστη μάλλον. Προσπαθήσαμε και στη δική μου χώρα και το κόμμα μου συμμετέχει στην κυβέρνηση. Είμαστε υπέρ των χαμηλών φόρων, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι απαιτούνται υψηλότεροι, τάξη, ε, υψηλότεροι φόροι, στοχευμένοι φόροι, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να κάνουν τις επιλογές τους. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε λύσει το θέμα. Το θέμα είναι να μπορούν οι πολίτες να διαλέγουν τον τρόπο κατανάλωσής τους. Και αυτό ισχύει και για τους κυρίους ε, Κορέι Αντεκάμπος και για την κυρία Μπαστός. Αναφερθήκατε και στις κοινωνικές συνέπειες και συμφωνώ. Αλλά η ανησυχία μου εδώ και ασχολούμαι με τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής πριν γίνω Ευρωβουλευτής, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις με κάποια τέλη ειδικά ή με κάποιους φόρους και να τα συνδυάσουμε και με άλλα κοινωνικά μέτρα. Αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό μόνο μέσω της τιμής της ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι και εγώ θα συμφωνήσω και θα καλυφθώ από αυτές τις ρυθμίσεις και αυτό δεν θα ήταν σωστό. Στην δική μου χώρα τουλάχιστον αυτά δείχνει η εμπειρία. Έχουμε ψηλούς φόρους και έχουμε ένα κράτος ε, κοινωνικών παροχών ισχυρών, κοινωνικής πρόνοιας ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι έχουμε ένα τέτοιο κράτος και προσπαθούμε να το τροφοδοτούμε. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρξει άμεση σύνδεση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε τον κοινωνικό τομέα. Δεν διαφωνώ λοιπόν μαζί σας. Και συμφωνούμε με την κυρία Ρούλε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για την κυρία Ρούλε βέβαια. Για μένα καλό είναι πάντως εντάξει. Χρειάζεται να πρασινίζω και λίγο κάπου κάπου. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπιέλλαν. Η Πολωνία είναι μια περίπλοκη περίπτωση. Υπάρχει μια χώρα που δεν δέχτηκε τον οδικό χάρτη και ήταν η δική σας. Είναι μια περίπλοκη χώρα. Είναι μια περίπλοκη χώρα. Είχα επισκεφθεί το 84 το, την Κρακοβία ήταν κίτρινη ατμόσφαιρα, θύμιζε το πώς ήταν το ρουργεμπίτ παλιά, ενώ τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Δεν ήταν ακριβώς μια περίληψη των λεχθέντων αυτό που κάνατε, αλλά είχε ενδιαφέρον. Για πρακτικά τώρα, για το πώς θα αξιοποιήσουμε σωστά την εργασία σας. Προθεσμία είναι η 5η Νοεμβρίου, 28 θα εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες, 29 θα ψηφίσουμε και θα ψηφιστεί και στην αρμόδια Κοιτάξτε, εγώ τις τελευταίες δύο μέρες του Οκτωβρίου θα είμαι στο Σουρινάμ με την αντιπροσωπεία ΑΚΕ. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να κάνετε μια αλλαγή. Είναι τόσο μακριά το Σουρινάμ. Θα το προσπαθήσουμε. Εξαρτάται και από το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Βιομηχανίας. Αν παραταθεί εκείνο μπορούμε να παρατείνουμε και εμείς το δικό μας. θα είστε ήδη στις 28 στο Σουρινάμα. Έχετε τόσα πολλά ενδιαφέροντα, κύριε Όλε Σμιτ. Δεν μπορούμε συνέχεια να σας έχουμε εδώ. Ευχαριστώ θερμά όλους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να περάσουμε στο τελευταίο μας ε, σημείο για σήμερα. Γνωμοδότηση και πάλι για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όμως που είναι καθήλια αρμόδια, αφορά τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μα είναι ο κύριος Χατζημαρκάκης, ε, ο κύριος Κορέντης ε, εκ των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Για το ΕΛΚ ποιος είναι σκιώδης, η κυρία Χάντσλικ. θερμή υπέρμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυρία Ρούλε είναι για τους πράσινους. Αν δεν είναι ο κύριος Μπιέλαν για τους μεταρρυθμιστές και, δημοκρα... και συντηρητικούς, θα κάνω εγώ τα σχόλια για την ομάδα. Δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί το σχέδιο γνωμοδότης. Μόλις ε, τώρα μοιράστηκαν, δεν κάνω προς το παρόν το είχαμε μόνο στα αγγλικά. Δεν έχουν λάβει όλοι τις μεταφράσεις, ε, κύριε Χατζημαρκάκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τώρα, εδώ κάνουμε λόγο για κάτι που 23 εκατομμύρια μικρο, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη αφορά δηλαδή την πρόσβαση στους χρηματοοικονομικούς πόρους, στα κονδύλια. Ξέρουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, νέων θέσεων εργασίας δημιουργήθηκαν από αυτές τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να πούμε και να διαπιστώσουμε ότι εξακολουθούν σε σχέση με την ευρωπαϊκή συμμετοχή εξακολουθεί ιδιαίτερα για την καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια Είμαστε υπανάπτυξη, εξακολουθούμε να είμαστε υπανάπτυκτοι. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση την οποία θεωρούμε ευπρόσδεκτη και χαιρετίζουμε ότι τα όσα υπάρχουν ως δράσεις ε, διαθέσιμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τα κράτη-μέλη πρέπει να συμπτυχθούν και να ενδυναμωθούν. Πολλά κονδύλια απαιτούνται να ξεκινήσει μια καινοτόμα επιχείρηση, καινοτόμος επιχείρηση και να προχωρήσει. Απαιτούνται τεράστια κονδύλια και αν διαφορετικές πολιτικές πολιτιστικές παραδόσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην Κίνα και στην Ασία από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν διαφορετικά αυτά τα προβλήματα. Είναι πιο ανοιχτοί στο πνεύμα τους για τέτοιου είδους ε, κινδύνους που επομίζονται και ξεκινούν μια τέτοια πορεία. Εμείς στην Ευρώπη δεν είμαστε τόσο ανοιχτοί. Το 7ο πρόγραμμα έρευνας και ε, καινοτομίας και είχα την τιμή να είμαι εισηγητής γι' αυτό όσον αφορά την εκπόνηση, την ε, δημιουργία αυτού του προγράμματος, τη γένεσή του. Ένα προϊόν το γνωρίζετε όλοι μέσω της ευρωπαϊκής αυτής προώθησης, ε, το οποίο είναι το κάλπ. Και μετά σταματάμε εκεί και ακολουθούν πολλά, πολλές επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο να περάσει προς τα έξω και έξω να γίνει ευδιάκριτο αυτό το, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Διότι πιθανότατα αυτή η μεγάλη επιτυχία των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν είναι τόσο γνωστή. Μετά η βελτίωση πρόσβαση σε κεφάλαια μέσα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Risk Shared Finance Facility, επιμερισμού κινδύνου ευρωπαϊκό μέσο και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν πολλά κονδύλια για την έρευνα σε καινοτόμε επιχειρήσει να διατεθούν με γοργότερε, ταχύτερε διαδικασίε και στον επιμερισμό κινδύνου ακριβώ περί αυτού πρόκειται, για την κάλυψη και αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Μάθαμε από του άλλου αυτό το μέσο το οποίο υφίσταται. Φαίνεται ότι υπόσχεται πάρα πολλά ε, στο μέλλον. Ιδιαίτερα για χώρες του Νότου ή που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση κονδύλια από το Ταμείο συνοχή ή από τα περιφερειακά ταμεία, να το Περιφερειακό ταμείο, ταμείο και Ταμείο ανάπτυξη να μπορέσουν να διατεθούν. Βελτιώνονται αυτά τα πλαίσια λοιπόν, ώστε εδώ καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τα προγράμματα Jessica, Jeremy να μπορέσουν υπό τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να οδηγήσουν σε αύξηση των κονδυλίων και πρόσβαση των κονδυλίων. Συνεχίζονται προγράμματα COSME, ορίζοντα 2020, όλα αυτά όμως πρέπει να διαπιστώσουμε και να πούμε ότι δεδομένων των μεγάλων αυτών επιβαρυντικών ε, συνοδευτικών ε, ε, δράσεων, ποια είναι αυτά, είναι η ενιαία εσωτερική αγορά. Θέλουμε καλύτερα να χρησιμοποιηθεί η ενιαία εσωτερική αγορά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγκρίναμε την Small Business Act. Όλα αυτά όμως μπορούν να λειτουργήσουν όταν θα έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, ένα υγιές σύστημα χρηματοπιστωτικής υποστήριξης. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δεν συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα από τα κυριότερα εγχειρήματά μας εδώ για τα όσα έχουμε εγκρίνει. Ιδιαίτερα η οδηγία περί ε, καθυστέρησης εξοφλήσεων λογαριασμών, Late Payment Directive. Ε, επενέσαμε ένα στον άλλο και είπαμε εγκρίθηκε αυτό επιτέλους. Γεγονός είναι ότι σε τέσσερα κράτη-μέλη η ηθική για αυτές τις πληρωμές είτε δεν είναι διαθέσιμη είτε δεν υφίσταται καν παρόλο τον κανονισμό μας ή δεν είναι καν διαθέσιμα κονδύλια. Ιδιαίτερα για κάποιες χώρες που πλήττουν με ε, ξεχωριστό τρόπο από την ε, κρίση αυτή, όπως ε, η χώρα για την οποία τόσο πολύ γίνεται λόγο σήμερα, η Ελλάδα για παράδειγμα, και καθυστερούνται εξοφλήσεις πληρωμών. Γι' αυτό δεν παραμένει τίποτα άλλο σε μένα ως συντάκτη γνωμοδότησης, σε εσά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι υποστηρίζουμε εσά για το πρόγραμμα δράσης το οποίο έχετε καταρτήσει, για το ότι θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί η πρόσβαση στα κονδύλια για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν θα φύγει μαγικά, δεν θα μπορέσει να αποβεί βάρος των, δεν θα πρέπει να αποβεί βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτή η κρίση. Το ευρωπαϊκό ε, σύστημα έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και σήμερα για έναν τέτοιο επιχειρηματία στην Ισπανία, ακόμα χειρότερα στην Ελλάδα, που προσπαθεί να βρει κάποια πίστοση, κάποιο δάνειο, δεν γίνεται, τίποτα δεν πάει. Έχουν κατεβάσει τα ρολά ε, τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό που πρέπει να προαχθεί σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται στις ε, χώρες που πλήττονται από την κρίση μπορούν, μπορούν οι άλλες χώρες να μάθουν πολλά πράγματα από αυτές. Έχουμε εδώ και το one stop shop, μία θηρίδα για όλους. Δηλαδή περί τίνος πρόκειται εδώ πάλι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στη χώρα τους φτάνουν στα όρια τους να μπορούν να αναζητήσουν δυνατότητες μέσω της μίας και ε, ενιαίας αυτής ρίδας, όπως σε άλλες χώρες ή όπως από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δοθεί μια τέτοια δυνατότητα πρόσβαση σε κονδύλια. Ηλεκτρονικά με πληροφόρηση μπορούν πάρα πολλά να επιτευχθούν. Θέλω να έρθω σε ένα θέμα το οποίο δεν διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στο πρόγραμμα πληροφόρησης. Όμως παρόλα αυτά είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή τράπεζες επενδύσεων ή τράπεζες ε, αρρωγής ε, που υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά όχι σε όλες. Εκεί όπου είναι γνωστές στη Γαλλία, για παράδειγμα κυρίως και στη Γερμανία, εκεί λειτουργούν καλά τα πράγματα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με πολύ καλό τρόπο κιόλα. Θα ευχόμαστε και θα ελπίζαμε να διεξαχθεί κάποια συζήτηση, να δούμε αν αυτά, παράδειγμα, τέτοιου είδους αρρωγές τράπεζες ε, όπως στη Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούσαν μήπως να δραστηριοποιηθούν σε άλλες χώρες. Διότι έχουμε εδώ ένα φραγμό πρέπει να πω θα μπορούσε να υποστηρίξει μια ξένη επιχείρηση, μια τέτοια ε, γερμανική τράπεζα αρρωγής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει όμως να προβληματιστούμε να δούμε αν θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον και υπό ποιου όρους. Διεξάγονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε σχέση με την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με πιο ενδυναμωμένο τρόπο στις χώρες που πλήττονται από την κρίση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να δοθούν μέθοδοι που να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που γνωρίζουμε από το Risk ε, ε, ε, Sharing Facility ή σε σχέση με το πρόγραμμα Jessica. Έχουμε την τεχνογνωσία. Πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε. Μπορούν να λειτουργήσουν αυτά. Εμείς ως Οικονομική Νομισματική Επιτροπή ΕΚΟΝ πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Κεφάλαια να διατεθούν σε, κάποια, σε κάποιες χώρες που αν μέσω του Περιφερειακού Ταμείου δεν αντληθούν, μέσω ενός τέτοιου μηχανισμού να μπορούν να εισρεύσουν στην οικονομία και κυρίως να καταλήξουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς όφελός τους. Να σας αναφέρω ένα αριθμητικό μέγεθος για την Ελλάδα που πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση. 40, 40% των κονδυλίων έχουν αντληθεί από αυτά τα κονδύλια. Όλα και όλα. Ένα χρόνο έχει ακόμα διάστημα τα 60% να μπορέσουν να κατανεμηθούν. Διαφορετικά θα ε, διαγραφούν αυτά τα κονδύλια για την Ελλάδα. Τώρα είναι επιτέλους η χρονική στιγμή. Μέχρι το, τέλος, μέχρι το 2013 ένα τέτοιο μέσο αρρωγής υποστήριξης να προχωρήσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συζήτησα και με τον, υπήρξε συζήτηση και με τον πρόεδρο Λάγκα και από πλευρά του κ. Χόγερ θέλει, ε, υπάρχει βούληση να προχωρήσουν. Ε, όμως έχω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ δεν πρόκειται για μεγάλα ε, προγράμματα και εγχειρήματα. Εδώ συγκεκριμένε δράσει δράσεις. 11 δι να μπορέσουν να διατεθούν όσο το δυνατόν πιο γοργά γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ποιότητα και πληροφόρηση. Επόμενο σημείο. Διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο. Rating, διαβάθμιση, βαθμολόγηση, θεμελιώδου σημασία. Παρόλη την οικονομική κρίση πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών να δίνουν σωστές πληροφορίες στις επιχειρήσεις σε, ε, στη, γλώσσα, σε, στη μία γλώσσα, στη γλώσσα που χρειάζονται. One stop shop, μία θηρίδα είναι η σωστότερη λύση. Γραφειοκρατία, επόμενο θέμα. Για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι μείζον πρόβλημα η, ε, η επαχθής κατάσταση όσον αφορά την γραφειοκρατική επιβάρηση και το χρονικό διάστημα που απαιτείται και τις υπογραφές και ε, άδειες στην Ελλάδα χρειάζεστε 20 υπογραφές για να, ιδρυθεί μια, να συγκροτηθεί μια νέα επιχείρηση. Υπερβολικά πολλές αυτές οι ε, υπογραφές και αυτές οι διεργασίες. Πάλι εδώ πρέπει να ασκηθεί επιρροή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μειωθεί αυτή η γραφειοκρατική επιβάρηση και να προχωρήσουμε σε ένα θετικότερο πλαίσιο. Για τις καθυστερημένες πληρωμές μίλησα, δεν είναι αποδεκτή η κατάσταση καθυστέρησης πληρωμών και πρέπει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα να αντιμετωπιστεί το δυνατόν ταχύτερα. Ένα επιπλέον ε, θέμα είναι το φορολογικό καθεστώς. Έχουμε διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και κυρίως ε, σε περίοδους κρίσης μέσω πίεσης της Τρόικας στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ενδεχόμενα στη συνέχεια αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε στην Ελλάδα που ισχύει αυτό τι είδαμε. Ζήσαμε μια αύξηση των φορολογικών επιπέδων της φορολογίας που το επίπεδο δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δυσχεραίνει τρομερά. Στην Πορτογαλία έχουμε και την παράδοξη κατάσταση αύξηση των φόρων να έχει έχει στραγγαλίσει την οικονομία με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει οπισθοδρομήσει, να έχει πάει πίσω σε σχέση με τα έσοδα, τα κρατικά έσοδα του κρατικού κορβανά. Τι καταδεικνύεται εδώ. Καταδεικνύεται ότι η πολιτική της Τρόικας ακριβώς χτυπάει, πλήτη αρνητικά τον ίδιο τον πυρήνα, την καρδιά της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ στην Πορτογαλία. Αυτό πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε και να διεξαχθεί μια συζήτηση για αυτό το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων, για παράδειγμα, Πρόεδρε, ώστε πιο, ε, με μεγαλύτερη σαφήνεια να αντιπαρατεθούμε με την πολιτική της Τρόικας. Πάνε πολλά πράγματα στραβά και αυτό δεν βαίνει καθόλου καλός και πρέπει να το ξαναδούμε. Ένα διαφανές πλαίσιο νομοθετικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα εμβαθύνω εδώ σε αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε και σε άλλα σημεία ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Να πω ότι καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες σε αγγλικά, σε αγγλική γλώσσα είναι πιεστικό αυτό ω προθεσμία. Είναι η 16 Οκτωβρίου. Εντάξει, αν θέλουμε να τηρήσουμε βέβαια το χρονοδιάγραμμα διάγραμμά Στις 5-6 Νοεμβρίου θα ξανασυναντηθούμε εδώ και θα τα εξετάσουμε τέλη Νοεμβρίου, 28-29 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε προς έγκριση. Ολοκλήρωσα, Πρόεδρε. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Well, thank you. Uh, Σας ευχαριστώ. Ε, σημείωσα αυτά που μας είπατε για τις ε, συζητήσεις που γίνονται στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Ε, γιατί οι πολιτικές που εξετάζονται εκεί έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομία. Από τους και ηγητές, πρώτα κυρία Χάντσλικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό ε, βέβαια υπάρχει τεράστια πολυμορφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ένα και μόνο τρόπο χρηματοδότησης για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, επαναλαμβάνω, τι ε, τις διαφορές, την πολυμορφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν και πολλές γνώσεις για τα οικονομικά και αυτό δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά τον οικονομικό τους προγραμματισμό και μπορεί να μπλοκάρει και την ίδια τους την ανάπτυξη. Και αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη, όπως μας είπε και ο εισηγητής, να δούμε πώς αυτή την κατάσταση θα τη βελτιώσουμε. Κατά τη γνώμη μου, θεμελιώδες είναι να γίνεται σωστός προγραμματισμός και των ε, σχεδίων των επιχειρηματικών ε, για να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις ώστε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια να μπορέσουν να τους εξασφαλίσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και όχι να τις επιβαρύνουν περισσότερο. Φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γιατί από αυτήν εξαρτάται και η ύπαρξη και η επιβίωση, αλλά και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότηση για, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Άνωση, αλλά εξαιτία τη άγνοια που έχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν μπορούν να αξιοποιήσουν όλου αυτού του μηχανισμού. Μια καλύτερη ενημέρωση λοιπόν για τι ευκαιρίε και τι δυνατότητε που έχουν για τη χρηματοδότηση οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι εξίσου σημαντικό θέμα και θα πρέπει και αυτό να το τονίσουμε. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πολύ σημαντικό είναι η άρση των φραγμών. Ιδιαίτερα του διοικητικού άχους και των διοικητικών εμποδίων. Ε, φυσικά ε, είναι δύσκολο να, για μια μικρή επιχείρηση να συγκεντρωθούν αυτές οι 20 υπογραφές και καλό θα είναι να πλουστευτεί η γραφειοκρατία και οι διοικητικέ διατυπώσει. Νομίζω ότι μια τέτοια απλούστευση θα διευκολύνει πραγματικά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για την πρόσβασή του στη χρηματοδότηση. Και φυσικά συμφωνώ και με το τελευταίο σχόλιο του κυρίου Συγητή. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι, ώστε η οδηγία για τις υπερήμερες πληρωμές να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στις εσωτερικές ένωμες τάξεις. Γιατί ακριβώ εξαιτία των καθυστερημένων πληρωμών πολλέ φορέ ε, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και μερικέ φορέ και την πτώχευση οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ζητώ συγγνώμη από του ε, υπόλοιπου συνομιλητέ, γιατί θα πρέπει να φύγω. Έχω στι 12.30 στο Voxbox ε, ένα ραντεβού. Ήδη έχω καθυστερήσει 20 λεπτά. Θα ήθελα πολύ να παραμείνω μέχρι το τέλο τη συζήτηση, αλλά πραγματικά αδυνατό. Αλλά θα ενημερωθώ για το περιεχόμενο τη συζήτηση και προσβλέπω σε πολύ καρποφόρα συνεργασία και με το εισηγητή και με του και εισηγητές. σα ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Σα ευχαριστώ πάντω που μείνατε μέχρι τώρα για να μα σχολιάσετε τι προσεγγίσεις. Είστε κι εσεί ιδιοκτήτρια α, περήφανη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε ξέρετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει από πρώτο χέρι. Ο κύριο Κορέντα Κάμπο. Ευχαριστώ Μάλκομ. Η γνωμοδότηση του κυρίου Χατζημαρκάκη είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πιο προχωρημένη από τις αρχικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι σχετικά άτολμες δεδομένες της σοβαρότητας της κατάστασης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι πραγματικά το πεζικό της παραγωγής ε, και της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι όλες ίσες, όπως μας είπε και η κυρία Χάντσλικ. Υπάρχει τεράστια πολυμορφία, μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συμβατικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν διατηρώντας τις θέσεις τους απασχόλησης και υπάρχουν και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται λιγότερο σε ό,τι αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί ε, οι, οι υπάλληλοι τους είναι πολύ νέοι και μόλις τελείωσαν τις σπουδές τους, αλλά έχουν προβλήματα πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση θα πρέπει να Τη συγχαίουμε, γιατί υπακούσε τελείω σε διαφορετικούς μηχανισμούς λειτουργίας και σε διαφορετικά συστήματα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε διαφοροποιημένη στρατηγική, παρόλο που με την παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση προσκρούσαμε σε κοινά εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο είναι το φορολογικό σύστημα. Και η υπερβολική εμπιστοσύνη ότι με την αύξηση του ΦΠΑ, στην Πορτογαλία για παράδειγμα, για τα εστιατόρια από 13% 23%, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αύξηση δικαιολογείται και ότι θα, προσθέσει, θα και μια άλλη αύξηση 1%. Παρ' όλα αυτά θα μειωθούν τα συνολικά έσοδα από το ΦΠΑ κατά 2% παρά τις διαδοχικές αυξήσεις που είχαμε. Βλέπετε λοιπόν ότι οδηγηθήκαμε σε παράδοξα αποτελέσματα για την υπερβολική εμπιστοσύνη που έχουμε στην αύξηση του ΦΠΑ. Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κοινό οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι το γραφειοκρατικό άχθο. Υπερβολικέ διοικητικέ διατυπώσει που επίση διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην Πορτογαλία μπορεί, θα μπορούσε κανεί να ιδρύσει μια επιχείρηση μέσα σε 20 λεπτά. Εξαιτία του Unstop Shop, τη μονοπευθυντική θηρίδα που ισχύει εδώ και 8 χρόνια. Είχαμε συγκεκριμένα σύστημα για να μπορεί κανείς ε, αμέσως να ιδρύει μια επιχείρηση. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στο κεφάλαιο, στα δάνεια από τράπεζες. Επίσης, ε, οι περίμενες πληρωμές του δημοσίου προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί ο αγοραστής, το δημόσιος αγοραστής δεν είναι επικίνδυνος επισφαλής αγοραστής, αλλά είναι υπερήμερος δυστυχώς αγοραστής. Αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις είναι εξίσου επικίνδυνος ένας υπερήμερος αγοραστής από ότι ένας αγοραστής πολύ μικρής εμβέλειας ή ένας ανύπαρκτος αγοραστής. Προσοχή λοιπόν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπερημέρες πληρωμές. Επίση, θα πρέπει να είναι πιο ευρηματική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προτάσει. Φυσικά συμφωνούμε με το One Stop Shop και αντίστοιχου μηχανισμού που ισχύουν στι διάφορε χώρε. Αλλά πιστεύω ότι εδώ έχουμε μία ευκαιρία ώστε στον κανονισμό για τι τράπεζε που τώρα εκπονείται, τώρα διαμορφώνεται μια τέτοια δομή για τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φροντίσουμε ώστε στον κανονισμό αυτό να υπάρχουν συγκεκριμένες προσα... κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι μεγάλες τράπεζες που λειτουργούν καλά ε, θα πρέπει να αρνούνται χρηματοδότηση στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί τα κεφάλαια που ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνήθω είναι και μικρά και μικρό διασυνοριακό αντίκτυπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι, οι τοπικές τράπεζες θα πρέπει να επιληφθούν αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πάντω τον εισηγητή τον κύριο Χατζημαρκάκη για την γνωμοδότησή του. Well, thank you very much. I know Mr. Rob is here from από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ο κύριος Ραμπ θα πάρει το λόγο, αλλά σαν σκιώδης και εγώ της δικής μου ομάδας να πω ότι πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο καλύπτει πάρα πολλούς τομείς δείχνει, υπογραμμίζει την περιπλοκότητα και την διαφορετικότητα των πηγών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων. Και γι' αυτό και μέσω του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου καλό θα είναι να εξηγηθούν όλες αυτές οι επιλογές που υπάρχουν. εξετάζει το σύνολο των μέσων τα οποία ταιριάζουν σε είδη επιχειρήσεων και στη φάση ανάπτυξή τους. Σωστά υπογραμμίζεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι, ε, οι μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις οι άγγελοι των επιχειρήσεων, οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κάποιο μέσο το οποίο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα από εταιρείε και στη δική μου εκλογική περιφέρεια όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα χρηματοδότησης. Συλλέγονται οι παλαιότερες εμπειρίες και βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες έτσι ώστε να καταστήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις τους ο συνδυασμός της εμπειρίας της χρηματοοικονομικής από τη μία και της διαχειριστικής από την άλλη είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και φορολογικά ευνοϊκά αυτοί οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο γιατί αναφέρθηκε και στο θέμα των δημοσίων προμηθειών. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ιδέες έτσι ώστε να τεθεί και το θέμα των καινοτόμων δημοσίων προμηθειών, γιατί έχουμε νέο μέσο στη διάθεσή μας για τις εταιρικέ καινοτομικές σχέσεις. Έχει σημασία οι χρηματοδότης να κατανοούν τη σημασία που έχουν αυτές οι δραστηριότητες γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία εργάζεται με έναν σημαντικό παράγοντα στον δημόσιο χώρο παραέχει εγγυήσει πολύ περισσότερες από ότι κάποια επιχείρηση η οποία δεν έχει αυτή τη διέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ενισχύσουμε και τον δημόσιο τομέα έτσι ώστε να αναγνωρίσουν ε, τους κινδύνους οι οποίοι θα είναι μικρότεροι στη συγκεκριμένη περίπτωση και έτσι τα χρηματοδοτικά μέσα να είναι ευκολότερα διαθέσιμα. Τώρα κύριε Ράμπα, ένα λεπτό. Ίσως να επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε μια διαφορετική φάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου για τη στήριξή σας και τα σχόλιά σας. Πράγματι το πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό στο πρόγραμμα δράσης μας περιλαμβάνουμε το σύνολο των πρωτοβουλειών τις οποίες θα αναλάβουν ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Υπάρχουν ε, πολλές επιχειρήσεις και πολλά είδη επιχειρήσεων και πολλά είδη ε, διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε ένα one-stop shop ε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές. Θα έχουμε επίσης μια ιστοσελίδα ειδική για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στον τομέα των καινοτομικών και στον τομέα διαφορετικών ταμείων και στον τομέα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διαφορετικού τύπου προγράμματα. Αυτό έχει σημασία και νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να ενημερώσουμε σωστά τις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενημέρωση επίσης είναι κάτι το κομβικό και στην περίπτωση της οδηγίας για τις πληρωμές με καθυστέρησης. Θα πρέπει να ενημερώνονται όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και τα δικαστικά σώματα και οι δικαστές γενικότερα που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν το Κοινοβούλιο για τη σημασία που δίνει σε αυτό. Παράλληλα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα διευκολύνουμε την πρόσβαση και να παρέχουμε περισσότερη χρηματοδότηση και στο μέλλον. Πράγματι έχουν υπάρξει επιτυχίες. Έχουν υπάρξει παραδείγματα λοιπόν επιμέρους ε, προγράμματα τοπικά και στη Γερμανία και στην Πολωνία και υπάρχουν επίσης ε, και κάποια application, κάποιες εφαρμογές οι οποίες ε, είναι πρωταγωνιστικές ε, στην χρήση του στα πλαίσια του iTunes, στη ζήτηση και έχουν χρηματοδοτηθεί από τα δικά μας προγράμματα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν σύντομα πάλι στον κύριο Χατζηματικάκη και μετά θα μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ για τις προτάσεις, συγκεκριμένες εξειδικευμένες προτάσεις, Μάκομ, και από πλευρά σου για το Business Angels ως θέμα τους αγγέλους των επιχειρήσεων. Με χαρά εγώ συντάκτης αυτής της γνωμοδότησης αν θα είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα από την Πορτογαλία, ιδιαίτερα όσον αφορά την φορολογική αυτή πτυχή τη αύξηση τη φορολόγηση, αν μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο πάντα λέγαμε και ω Ευρωκοινοβούλιο, ότι η ψηλότερη φορολογία δεν οδηγεί στο να πάει καλύτερα η οικονομία. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αγαπητέ Μάκομ, συμβαίνει το εξή. Μια εβδομάδα θα έχουμε όλοι και όλοι για τι τροπολογίε. Γι' αυτό βρισκόμαστε υποπίεση 5-6 Νοεμβρίου σε, θα ξανασυναντηθούμε και θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 27-28 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ Μάκο. Well, I know that it's a tight timetable um, I'm sorry that... Uh, Πιεστικό το χρονοδιάγραμμα, το γνωρίζω. Λυπούμε που δεν είχαμε έγκαιρα τις ε, εκθέσεις για αυτή τη συνεδρίαση. Θα είναι διαθέσιμες υστερότερα, αργότερα αλλά για να τα καταφέρουμε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ε, συνάδελφοι υποβάλλουν τροπολογίες στα αγγλικά και αυτό θα ήταν επικοδομητικό. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλα αυτά και σίγουρα θα δούμε τα θέματα αυτά στις τροπολογίες. Πρωτού κλείσουμε τη συνεδρίαση να υπενθυμίσω σε όλους ε, για άλλη μια φορά ότι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα την εβδομάδα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ξέρω ότι θα έχετε εκδηλώσει στις χώρες σας πολλοί από εσά. Και την εκκίνηση, καθέλκυση τη Δευτέρα συνολικά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσβλέπω ώστε να σας ξανασυναντήσω. Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα ξανασυναντηθούμε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα 15.00. Θα έχουμε δύο συνεδριάσεις την 3η 6 Νοεμβρίου στις 9 και στις 3 9 το πρωί και 3 το απόγευμα. Θα σας ξανασυναντήσω τότε. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Λίγη συνεδρίαση. Γεια.